Good afternoon to everybody and I... Καλησπέρα. Ελπίζω να είχατε ένα χαλαρωτικό υγιές γεύμα για να αντέξετε μέχρι τις 6.30. Έχουμε πολλές αναφορές. Ελπίζω να είμαστε αποτελεσματικοί. Κάτι που θα είμαστε αν το προσπαθήσουμε όλοι. όντας συνοπτική και ακριβής. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών, εγκρίθηκε η... το πρόγραμμα για τον Οκτώβριο μαζί με τη 1307 και το 1073 ξανά Δεν υπήρξε κάποια ένσταση, δεν υπήρξε ανάθεση εκθέσεων και έπειτα είδαμε τα σημεία Β όπου εκεί έχουμε κάποιες υποθέσεις οποίες θα κλείσουμε γιατί δεν είχαμε πάρει πληροφορίες για την 884 και 900 τις κρατάμε ανοιχτέ, γιατί είχαμε παραπάνω πληροφορίες μας έδωσαν οι αναφέροντες για τις ε, επισκέψεις μας, τη διερμητική επίσκεψη στη Λάρνακα συγκεκριμένα έχουμε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα Προσωπικά δεν θα λάβω μέρος στην αντιπροσωπεία. Ευτυχώς όμως έχουμε τον νέο πρόεδρο, τον Παλ Τσάκη, τον νέο επικεφαλής αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Οι συντονιστές επίσης ε, έλαβαν απόφαση ή θα λάβουν απόφαση για τα διάφορα hearing στις 11 Οκτωβρίου και θα έχουμε και μία ακρόαση για την επισφαλή απασχόληση 22 Νοεμβρίου. Θα πρέπει να στείλουν οι ομάδες προτάσεις τους πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα συνδυάσεων για το 2018 εγκρίθηκε και σε συνέχεια στην αναφορά 447 θα διοργανωθεί ένα εργαστήριο που θα ζητήσουμε να το διοργανώσει το θέμα τικό τμήμα Γ. Το EFTD ζήτησε μετάφραση της έκθεσης της ομάδας εργασίας ε, για την ε, δεξιά των παιδιών εγκρίθηκε και θα ζητηθεί παρέκκληση από εμένα προς τον προ. Επίσης, ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων είχαν οι συντονιστές για το παραδεκτό των τροπολογιών στην Επιτροπή μας. Φυσικά και βοηθάει να αναφερόμαστε στις φυστάμενες αναφορές ως τεκμηρίως των τροπολογιών. Αλλά αυτό δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για να κρυθούν παραδεκτές τροπολογίες. Επίσης επικαιροποιήθηκε ε, η πύλη πέτη και ακούσατε τα σχετικά, οι συντονιστές και υπήρξε και ενημέρωση για μια σειρά από έγγραφα. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι το πρωί ολοκληρώσατε την έκθεση για την ε, ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει οι ομιλητές. Ο κ. Μαριάς, λοιπόν. Πέδρε, ε, πράγματι δεν είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε στο report. Θα είμαι σύντομος. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε την έκθεση για την ε, European Citizenship του 2017 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια όπως ε, ερμηνεύεται στα ελληνικά. Α, όταν είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο το 1993 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είχαμε την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης να συζητήσουμε αρκετά θέματα γύρω από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και είχαμε επικεντρωθεί οπωσδήποτε στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ως πολιτικό δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαφορετικό από το οικονομικό δικαίωμα να εργάζεται και να κυκλοφορεί ελεύθερα. Επίσης είχαμε αναφερθεί στο δικαίωμα αναφοράς, ένα δικαίωμα το οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι ασκείται σημαντικά εδώ σε αυτή την ε, Επιτροπή. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση σημαντικά αναφέρεται στα θέματα αυτά. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, ένα γεγονός που πιστεύω ότι απασχολεί χιλιάδες πολίτες, απασχολεί και χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν αναγκαστεί λόγω της Τρόικας και της μνημονιακής επίθεσης που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα να φύγουν από τη χώρα μας, να μεταναστεύσουν και πάρα πολλοί από αυτούς νέοι επιστήμονες κυρίως βρίσκονται στην ε, Βρετανία. Ε, το σημείο που με ενδιαφέρει να θίξω είναι το σημείο 10 και έχει σχέση και με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Διότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι μια αρμοδιότητα καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που βεβαίως οι νομοθεσίες των κρατών μελών μπορούν να τις συμπληρώνουν όμως δεν μπορούν να είναι τέτοιες οι νομοθεσίες των εθνικών κρατών που να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήθελα να αναφέρω ότι στην Ελλάδα ο νόμος ο οποίος ε, πέρασε προκειμένου να είμαστε υποψήφοι ευρωβουλευτές είναι αντίθετος με το κοινοτικό δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υποχρεώνει τους βουλευτές οι οποίοι είναι εν ενεργεία να παρετηθούν προκειμένου να είναι υποψήφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και στη Λάτβια. Θεωρώ ότι είναι αντίθετο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχα πει τότε όταν ήμουν βουλευτής. Εγώ αναγκάστηκα να παρετηθώ από βουλευτής μαζί με ορισμένους άλλους συναδέλφους και βεβαίως δεν γνωρίζαμε αν θα εκλεγούμε ή όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε όλα τα άλλα κράτη υπάρχει το ασυμβίβαστο. Δηλαδή κατεβαίνει στι εκλογέ και από εκεί και πέρα αν εκλεγεί Ευρωβουλευτή επιλέγει αν θα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή θα παραμείνει στην Ελληνική Βουλή. Ο ελληνικό νόμο επιβάλλει κόλλημα. Κόλλημα υποψηφιότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Και ένα δεύτερο θέμα και τελειώνω είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών στην δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς ως ευρωβουλευτές να εκφράσουμε τις απόψεις μας εκπροσωπώντας και τις πολιτικές μας ομάδες και κυρίως να έχουμε τη δυνατότητα οι απόψεις αυτές να εκφράζονται και να κοινοποιούνται στον ελληνικό λαό. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση τουλάχιστον απέναντι σε μένα ως βουλευτή, ως ευρωβουλευτή και μέρος του ECR. Υπάρχει συστηματικός αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που σας λέω το έχω καταγγείλει δύο φορές στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η κρατική τηλεόραση στο Στρασβούργο που έρχεται μια φορά το μήνα να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διοργανώνει εκπομπές όπου συμμετέχουν τρεις συνάδελφοι εκπρόσωποι Φερρυπίν της ΓΚΟΕ, ένας της, ε, του, του EPP, ένας της Σοσιαλιστικής Ομάδας και κανένας του, του ECR. Αυτό είναι απαράδεκτο, το έχω καταγγείλει και θα πρέπει κάτι να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Μας αποκλείουν συστηματικά και έχουμε όλα τα στοιχεία από τις κεντρικές εκπομπές που γίνονται όχι μόνο στην κρατική τηλεόραση αλλά και στα υποτιθέμενα μεγάλα κανάλια. Άρα λοιπόν κλείνω και θα βάλω μια τροπολογία στα θέματα αυτά για να υπάρξει δημοκρατικός διάλογος και συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει οι πολιτικές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους στα κράτη-μέλη και υπάρχει υποχρέωση πλουραλισμού Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα κράτη οφείλουν με αντικειμενικότητα να παρουσιάζουν όλες τις απόψεις. Και όσον αφορά το ECR και εμένα προσωπικά υπάρχει συστηματικός αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα που θέσατε. Ίσως όμως έπρεπε να τα πείτε στην ε, διοίκηση του Κοινοβουλίου, γιατί δεν έχει και καμία μεγάλη σχέση με την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που συζητούμε. Πάντως ε, θα σας παρότρινα να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες για αυτά που μας αναφέρατε. Η κυρία Στανόκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πολύ καλό το κείμενο της Μπεατρίθ. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αναφέρεται στο Brexit μεταξύ άλλων. Και αναφέρεται στα προβλήματα ιδίως των ατόμων που έχουν μετακινηθεί, από, μετεγκατασταθεί από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο και τώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και αυτό αφορά και τους Βρετανούς υπηκός που ζουν στα κράτη-μέλη της Υπηρετικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τούμπαλιν. Υπάρχει ένα ψήφισμα που τη γνωρίζω το οποίο έχει εκπονήσει η διαπραγματευτική ομάδα για τον Brexit και θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στο Λομέλη. Δεν ξέρω αν καλό θα ήταν να περιλάβετε τις προτάσεις μας όχι μόνο στις ετολικές σκέψεις αλλά και στο σώμα της έκθεσης, δηλαδή ότι τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων είτε Βρετανών επικών που ζουν στην υπόλοιπη Ένωση, είτε των Ευρωπαίων επικών που ζουν στη Βρετανία, να μην πληγούν. Πρέπει να θέλουμε να αναφέρεται στο σώμα της έκθεσης. Σε ό,τι αφορά το εργαστήριο, υπάρχουν ε, ε, για την ιστονία, από την Εστονία και τη κάποιες αναφορές για τα λογικά τους δικαιώματα και αντίστοιχα περιπτώσεις από τη μια χώρα της Σοβιετικής δημοκρατίας λέει η πρόεδρος στην άλλη. Υπήρξαν ε, μετακινήσεις τέτοιες, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή χάσανε τα δικαιώματα οι πολίτες του εκλέγει και εκλέγεστε. Και υπάρχει για ένα ιδιαίτερο καθεστώς που τους ε, αφορά. Ότι δηλαδή υπάγονται στη Λιτωνία και στην Εστονία γιατί ουσιαστικά δεν έχουν ε, την ε, ηθαγένεια κάποιου κράτους. Θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβουμε και αυτούς τους ανθρώπους όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Έχω κάποιες τροπολογίες που θα καταθέσω. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Είναι εξαιρετική η έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εύη, είστε και εσείς Θέλετε το λόγο. Σεσίλια, σε ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Μπράβο και από μένα για τη δουλειά της συναδελφού Μπεθέρα. Εάν κανείς θέλει εδώ να περιοριστεί στην ε, ρητορική μιλώντας για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια ε, τότε θα έπρεπε να περιοριστεί στη, στο βυτικό επίπεδο, σε κάποια δικαιώματα αλλά το θέμα είναι και τι γίνεται από ηλικής πλευράς πρακτικής για τους Ευρωπαίους και συμφωνώ με τις επικρίσεις του σχεδίου κειμένου και εκεί διατυπώνει επιφυλάξεις, αμφιβολίες σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανησυχίες και τα προβλήματα των πολιτών και σίγουρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προσπαθήσει κανείς και να ζυγίσει, να αξιολογήσει αυτό, αυτή την έννοια, την ηθαγένεια, την ευρωπαϊκή και κατόπιν να δούμε τι ισχύει στους διάφορους τομείς, περιβάλλον, υγεία κλπ. και από πλευρά κοινωνική δικαιοσύνη. Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να μπορέσουμε να καλύψουμε και να αξιοποιήσουμε την έννοια της ηθαγένειας που πάει χέρι-χέρι με την εθνική, ας πούμε, ηθαγένεια. Έτσι θα υπάρξει πρώτη στη θέμενη αξία. Συμφωνώ 100% για τις επικρίσεις του κειμένου που αφορούν αυτή την απίστευτη καθυστέρηση της οδηγίας κατά των δεσμενών διακρίσεων. Την περιμένουμε σχεδόν 10 χρόνια. Τέλος. Πιστεύω ότι χρειάζεται εκ βάθρων να αναθεωρηθεί το σύστημα διακυβέρνησης. Να υπάρξει διαφάνεια. και έτσι να έχουμε πρόοδο σε όλους τους τομείς, σε όλα τα μέτωπα. Και επήγε επομένω το να εγκαταλείψουμε τον μερκαντιλισμό και τη λιτότητα που τώρα χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Και πάλι ευχαριστώ συνάδελφα και θα κατεβάσω κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λέει η κυρία Τώρα η Μαρία Λεμπουλόζη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια για την Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Τι καταδεικνύεται η δέσμευση της Ευρώπης. Όλα τα θεσμικά όργανα συμφωνούν γιατί πρέπει να προχωρήσουν προς αυτό το μέτωπο αλλά και τα κράτη-μέλη. Θυμάστε πέρσι το Μάρτιο ότι κάναμε, κάναμε εκείνη την ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μαζί με τη Γιούρη σε συνεργασία και με την ΑΦΚΟ και την ΛΥΜΠΕ το οποίο συνέβαλε πολύ στην έκθεση αυτή. Καθορίσαμε τις προτεραιότητες, αποφασίσαμε για δράσεις ούτως ώστε να αξιοποιηθούν τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, τα καθημερινά δικαιώματα για την καθημερινή ζωή, για να υλοποιήσουμε τις κοινέ αξίες και την δημοκρατική συμμετοχή. Ευχαριστούμε για τις ιδέες που εισφέρει η έκθεση. Έτσι θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα με τις προτεραιότητες τους να καλύπτουν τα προβλήματα των πολιτών. Υπενθυμίζω όμω ότι πρόκειται για δέσμη μέτρων. Εν προκειμένου έχουμε αυτή την έκθεση με τι προτεραιότητε, αλλά παράλληλα έχουμε και μια άλλη έκθεση που έχει με το άρθρο 25 της συνθήκης. Το τι έγινε την τελευταία τριετία και τι θα γίνει στο μέλλον. Βλέπουμε επίση πώ υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσει του παρελθόντο και τι έγινε με τι παλιότερε προτεραιότητε. Μια που πιέζει ο πρέπει να σα πω ότι έχουμε πολλέ προτεραιότητες που αναφέρονται στην έκθεση και μία από αυτές είναι ότι θα γίνει μια ενημερωτική εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη πριν τι ευρωεκλογέ για τα δικαιώματα που συνδέονται με την Χρειάζεται να ενημερωθεί ο κόσμος για τα δικαιώματα τους και την άσκηση αυτών. Εδώ καθορίζονται κάποιε δράσει και κάποιε προτεραιότητε για δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Διάφορε πρωτοβουλίε για τι αριστερέ πρακτικέ, για τα δικαιώματα τα σχετικά με τι εκλογέ, που είναι πολύ σημαντικά. Άλλο σημαντικό, με κάποια άλλη δράση θέλουμε να πλουστεύσουμε, να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή. Και πρόσφατα ξέρετε ότι είχαμε κάποιε προτάσει για την νέα ψηφιακή πύλη για να βοηθήσει επίσης τα διασυνοριακά δικαιώματα. Και η ισότητα βέβαια έχει πρωταγωνιστική θέση σε αυτά. Αναφερθήκε σχετική οδηγία. Είναι προτεραιότητα της Επιτροπής σας. Ήταν αυτά και στις κατευθυντήριες του Πρόεδρου Γιούγκερ. Έχει δεσμευτεί η Κομισιόν επομένως. Επίσης, εξονίζουμε τις διατάξεις σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, σχετικά με την προξενική προστασία, ταυτότητες, έγγραφα σχετικά με την νόμιμη κατοικία. Και χτε δημοσιοποιήθηκαν κάποια σχετικά στοιχεία. Εδώ βάζετε λίγα γιατί ξέρω δεν έχετε χρόνο και αν υπάρχουν ερωτήσει να τι απαντήσω. Ευχαρίστω. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα είναι ενδιαφέρον να ακούμε τις παρατηρήσεις σας. Ζήτω συγγνώμη που ε, χρειάζεται να σας διακόψω, πρέπει όμως να προχωρήσουν. Θα ήθελα να δω αν είναι παρόν ο κύριος Δεν είναι. Να δώσω το λόγο λοιπόν πάλι στην κυρία Μπεθέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δράτω με της ευκαιρίας και θα χρειαστώ μόνο ένα λεπτό γιατί το μόνο που θέλω να κάνω ουσιαστικά είναι να ευχαριστήσω θερμά όλου του συναδέλφους που θα συνεργαστούν μαζί μου και τους Κιώδης και όλους τους υπόλοιπου συναδέλφους που θα συνεισφέρουν σε αυτή την έκθεση, διότι έχουμε μία δέσμευση. Πρέπει να έχουμε κοινού στόχου, να είμαστε σαφείς και αποφασισμένοι. Και ο συγητή ε, από τη ΛΥΜΠΕ συνεργάζεται και όλοι οι συντάκτες ονομοδότηση. το ίδιο. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Μπουλανζέ και για τη δουλειά της και για την καλή της διάθεση. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή ε, και έχουμε συζητήσει ώστε να υπάρχει σύγκληση απόψεων. Και ξέρουμε ότι έχουμε έναν κοινό ενίο στόχο. Ότι δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα πρέπει να εργαστούν ευθυγραμμισμένα και ενωμένα για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η οποία βασίζεται σε τρει πυλώνες. Την ισότητα που σημαίνει καμία διάκριση, το δικαίωμα υποβολή αναφορών και τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα τα άλλα είναι σε δεύτερο πλάνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον οικοδομητικό, διαφωτιστικό αυτό τρόπο και μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου θα περιμένω τις τροπολογίες σας. Ελπίζω να έχουμε και στις 22 Νευρίου που θα ψηφίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όπως είπαμε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 28 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα πραγματοποιηθεί 22 Νοεμβρίου. Μια υπενθύμηση για όσους από εμά βρεθήκαμε στον Τάραντα στην Ιταλία. Ε, πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα θα υπάρχουν στην τελική έκθεση που προβλέπεται για τέλη Οκτωβρίου. Θα ήθελα όμως να σας αναφέρω τι συμφώνησαν όλοι στην αποστολή. Και για την... Ε, είναι, είναι λοιπόν απαραίτητη η ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον ε, για τους ανθρώπους της περιοχής. Δηλαδή, διάλογος ανάμεσα στην ε, ηγεσία των επιχειρήσεων και τους πολίτες. Ε, αυτό συμφωνήθηκε από όλες ε, τις πλευρές. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα στον τομέα αυτών. Ως πρόεδρος της αποστολής στην συνέντευξη τύπου μετά από την αποστολή αυτή είπα και σας επαναλαμβάνω σήμερα ότι στο πνεύμα της σύμβασης του όρχους απαιτείται πιο συμμετοχική προσέγγιση απέναντι στους πολίτες που θα βοηθήσει να επανοικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των κύκλων συμφενόντων της περιοχής αυτής. Αυτό έλειπε. Χωρίς ε, να θέλω να ε, γεννήσω μεγάλες προσδοκίες για την έκθεση, αυτό έχουμε να πούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, το σημείο 16 έχει αναβληθεί. Έχουμε λοιπόν τώρα την ε, αναφορά 0867 κάθετος 2016 που είναι το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Απαγόρευση χημικών και βαρέων μετάλλων ε, στα παιδικά παιχνίδια. Ε, φαίνεται τρελό το να πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Ε, δίνω λοιπόν το λόγο κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθότι ο αναφέρον δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Κύριε Φόγγελσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία για τα παιχνίδια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει πολύ αυστηρές διατάξεις σχετικά με τα χημικά και τα βαρέα μέταλλα στα παιχνίδια. Ε, τα όρια έχουν τεθεί με τέτοιο τρόπο που μόνο το 10% της ασφαλούς ποσότητας ε, επιτρέπεται ε, να περιέχονται στα παιχνίδια για τα χημικά και για τον μόλιδο και τα ε, και για τα βαρέα μέταλλα το ποσοστό αυτό είναι 5%. Έτσι υπάρχει περιθώριο για επικίνδυνες ουσίες από άλλες πηγές. Έχει γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία επίσης για το μόλιβδο και το κάδμιο. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ αυστηρά, αυστηρούς κανόνες. Επίσης για τη δυσφενόλη α έχουμε πολύ αυστηρό όριο και πρόσφατα. Ε, το όριο αυτό ε, έγινε πιο αυστηρό κατά 2,5 ε, φορές. Το 2009 υιοθετήθηκε η οδηγία αυτή, έκτοτε έχουν γίνει πιο αυστηρά τα όρια 10 φορές, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επιστήμης. Διότι θέλουμε έτσι να προστατεύσουμε τα παιδιά από πιθανούς κινδύνους. Θα ήθελα να προσθέσω όσον αφορά την δεύτερη αυτή αναφορά για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου τα κράτη-μέλη είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των ε, παιχνιδιών. Θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια ε, χρηματοδοτεί σχετικές ενέργειες. Ο έλεγχος ε, των παιχνιδιών παίζει σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος και τώρα οι συνάδελφοι έχουν λόγο think we Οπότε θα μπορούσαμε να καταλήξουμε οριστικά σε σχέση με αυτή την αναφορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπαινθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προς ενημέρωση αυτή η αναφορά γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει κάποιο είδους ε, πρόταση ε, για την απαγόρευση αυτών των χημικών. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια ξέρει την απάντηση. Διότι έχουμε αυτές τις χημικές ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και είναι αιτία προβλημάτων ε, αναπαραγωγικών και ενδοκρινικών διαταραχών. Οπότε να ενημερώσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντο. και να στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσουμε εάν υπάρχει κάποια πρόταση για απαγόρευση, ε, πρόθεση απαγόρευση των αυτών των χημικών και να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Εντάξει. Τέλεια, σας ευχαριστώ. And we move to the next petition, which is... Μέτρα στην επόμενη αναφορά είναι η 30. Προέρχεται από τον Ολιβιέ Μπαρτέλ και αφορά τους πλαστικοποιητές σε αντικείμενα καθημερινή χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εδώ ο εισηγητή. And I'm happy to extend the Η εκπρόσωπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιοδήποτε εξημών μπορεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέρον ζητεί να απαγορευτεί η χρήση αυτών των πλαστικοποιητών, συγκεκριμένα των φθαλικών ενώσεων που περιέχουν τους πλαστικοποιητές να μην χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα καθημερινές κρίση. Η απάντησή μας βεβάστηκε τον Μάρτιο του 2016. Από τότε έχει σημειωθεί πρόοδος στους αφορά αυτές τις ουσίες. Να σας παρουσιάσω τι περιέχει το πιο πρόσφατο εγγραφό μας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΕΚΑ για τη Δανία που περιέχονται όλα αυτά στο έγγραφό μας του Μαρτίου και η ΕΚΑ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της σχετικής πρότασης. Ελέγχθη ότι υπάρχει όντως κινδύνος για την υγεία και ότι θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση αυτών των ε, χημικών ουσιών. Υπήρχε μια μεταβολή στη γνωμοδότηση στις 29 Αυγούστου, πολύ πρόσφατα δηλαδή. Και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον κανονισμό REACH, τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προπαρασκευάσει μια πρόταση για την απαγόρευση αυτών των ε, ουσιών από τα καθημερινά αντικείμενα. Και θα διαβάσουμε όπου πρέπει, σε κράτη-μέλη, ρίτς κλπ τέλη του, του έτους. Τώρα, έχουμε τέσσερα άρθρα για τις αντίστοιχες φθαλικές ενώσεις, DHP, DVP, DVP, EBP. Πρόκειται για τις ουσίες με τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει καθημερινή επαφή μέσω μεμβρανών, μέσω εισπνοής, μέσω επαφής ε, από αυτά τα αντικείμενα καθημερινής χρήση εσωτερικού χώρου. Οπότε η απαγόρευση μπορεί να καλύψει επίση την άμεση έκθεση για κάποια αντικείμενα τα οποία ε, μπορεί να έρθουμε σε επαφή σε χώρους. Ας πούμε στον κήπο. Έτσι νομίζω θα συμπληρωθεί η απαγόρευση που όπω είπαμε ήδη υπάρχει, ανέφερε η πρόεδρος προηγουμένως για της Αυθαλικές Ενώσης στα παιχνίδια. Ήδη υπάρχει αγόραση για τα παιχνίδια και για άλλα αντικείμενα που σχέση με τους ανηλίκους. Είπαμε οπότε ότι άλλαξε τώρα η λίστα των παραμένων ουσιών σε κάποιες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Και έτσι καλύπτονται και αυτές οι τέσσερις θαλικές ενώσεις και αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή η υπογόρευση του 2019 τέλος. Συνεπία της πρόσφατης νομοδότησης της ΕΚΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την ΕΦΣΑ την εταιρεία ιδιοδοτική ασφάλεια να αναθεωρήσει τη γνωμοδότηση του 2015 που ε, αφορά τα DEHP φθαλικά όσον αφορά ε, κάποια πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα οπότε θα ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση και εμείς θα αποφασίσουμε τι μέτρα θα λάβουμε για αυτά τα υλικά που έχουν συμπαθεί με τα είδη διατροφής. Άρα θα κάνουμε όλες αυτές τις ε, δράσεις και ενέργειες ούτως ώστε να περιοριστεί η χρήση αυτών των φθαλικών όπως ζητεί ο αναφέρον. Thank you much. Floor is open for colleagues. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Ελεονόρα. Sì, grazie Presidente. Eh, io vorrei capire... Θα ήθελα να καταλάβω, Πρόεδρε, καλύτερα το εξή. Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα αυτή η ενδοκρινική διαταράκτηση αυτών των ουσιών είναι κάτι το οποίο έχει διευκρινιστεί και ξεκαθαριστεί. Όταν όμως γίνεται αυτή η αναφορά στην, στον περιορισμό στη χρήση αυτών των ενώσεων στα αντικείμενα καθημερινής χρήση. Ελπίζω ότι αυτό σημαίνει πλήρη απαγόρευση χρήσης. Άλλωστε υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικέ. Θέλω να με διαβεβαιώσει προς το Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σας παραπέμπω και στο Refit. Να μην ανοιχτεί η αναφορά σας προτείνω και να την ε, κοινοποιήσουμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Nobody Δεν ζήτησε κανείς άλλο το λόγο. Καθότι γνωρίζουμε ότι η οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015 και θα ισχύσει από το 2019, Στο μεταξύ μπορεί να υποβληθούν αιτήματα για παρεκκλήσεις από την ε, σχετική βιομηχανία. Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε εάν θα επιτραπούν και θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εξέταση αυτών των παρεκκλήσεων για να δούμε εάν θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή εάν θα πάψουν να ισχύουν. Αυτό λοιπόν θα ήταν χρήσιμο. Μήπως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει με τη σχετική περιγραφή και επίσης ε, να μας ε, περιγράψει μελλοντικά μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Στο μεταξύ θα ήταν χρήσιμο, όπως είπε και η Ελεονόρα, να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να λάβουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτός. Συμφωνείτε. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιτροπή ΕΝΔΙ και να ζητήσουμε την γνωμοδότησή τους. Συμφωνείτε? Χρειάζεται να επιδείξουμε συνέπεια. Νομίζω ότι όταν υπάρχει οδηγία την οποία καταφέραμε να υπερψηφίσουμε μετά από πολλή πίεση και μετά από πολύ, πολύ πολιτικό διάλογο, δεν θα πρέπει απλά να εγκαταλείπουμε τα πράγματα όταν τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στα παρασκήνια, εφόσον είναι δυνατόν. Συμφωνείτε, βλέπω ότι οι συνάδελφοι γνέφουν καταφατικά. Το ΕΛΚ σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε τώρα στην αναφορά 2341 για τη βυσφενόλη Α. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον, είναι όμως ο Τζόναθαν Πρίζα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το 2013 ο αναφέρον ζητούσε απαγόρευση της χρήσης της δυσπενόλης α στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας επικαιροποιήσω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014. Η ΕΦΣΑ έχει δημοσιεύσει πλήρη γνωμοδότηση το 2015 σχετικά με τους κινδύνους της δυσφενόλης α, BPA, ε. στα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνέπειες, μεταξύ άλλων ε, τις ενδοκρινολογικές διαταραχές. Και έχει ε, καθορίσει ένα ασφαλές όριο για την πρόσληψη της ουσίας αυτής. Επίσης υπήρξαν πρόσθετες ε, έρευνες ε, της ΕΦΣΑ πέρσι το 2016 που δεν ε, οδήγησαν σε τροποποίηση του συμπεράσματος της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε στα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ και έχει μειώσει κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια της δυσφενόλης Α και σκοπεύει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής ε, ε, πέρα από τα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Υπάρχει κάποια επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυσφενόλη α ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευάλωτες ηλικιακές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ενισχύσει το μέτρο για προστασία των βρεφών και των μικρών παιδιών μέχρι την ηλικία των τριών ετών, προτείνοντας ε, απαγόρευση ε, για την ε, μεταφορά της δυσφενόλης α στα τρόφιμα από άλλα υλικά. αναμένονται νέα δεδομένα και νέες ε, έρευνες ε, σχετικά με τις αβεβαιότητες αυτές. Όσον αφορά τη χρήση της δυσφενόλης α σε άλλα προϊόντα, τροφή, ε, σε άλλα προϊόντα, έχουν εφαρμοστεί νέα όρια για τα παιχνίδια που θα ισχύσουν από του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει υιοθετήσει κανονισμό για την χρήση της δυσφενόλης α σε θερμικό χαρτί που συνήθως χρησιμοποιείται για αποδείξεις καταστημάτων. Επίσης, εμπίπτει στον κανονισμό REACH λόγω των ε, ενδοκρινολογικών διαταραχών που μπορεί να προκαλέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε, η γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ήταν του 2014, οπότε ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε εδώ. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι, εφόσον θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω να στάει κανείς το λόγο. Εγώ προτείνω να κάνουμε το εξής, διότι είχαμε τώρα πλήρη επικαιροποίηση ε, πλήρη ενημέρωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την αναφορά αυτή, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μια σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Συμφωνείτε? Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ. Και προχωράμε στην επόμενη αναφορά, υπαριθμών 1075, ε, σχετικά με τις εικαζόμενες βλάβες που προκαλούν τα αποσμητικά χώρου. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, είναι όμως παρόν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνω το λόγο στην Άννα Μαρία Μπλάς Ρίκο ή την Βαλεντίνα Μπερτάτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις χημικών ουσιών που βρίσκονται σε αποσμετικά χώρου για τους καταναλωτές ε, και ιδίως ε, για τις ε, εκπομπές από τα Συγγνώμη, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω τι ακούω. Είναι μια γλώσσα άγνωστη στα ακουστικά μου. As well. Um, you want me to speak in English? Θέλετε να τα πω αγγλικά μήπως? Όχι με το ζόρι, λέει ο πρόεδρο. Νομίζω ότι εντάξει, λειτουργεί η αγγλική καμπίνα. Ενδιαφέρον αυτό που συνέβη. Ωραία, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα λοιπόν, εφόσον μου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο αναφέρον εκφράζει τις ανησυχίες του για τις αντικέ επιπτώσεις ε, των χημικών ουσιών ε, σε διάφορα ε, προϊόντα καθημερινής χρήσης, τους καταναλωτές και ιδίως εκπομπές από τα κοσμητικά χώρου και αναφέρεται σε μία μελέτη του 2005 και στην εκ αξιολόγηση επιστημονικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες μελέτες που έχουν γίνει για τα προϊόντα αυτά, ε, μεταγενέστερες μελέτες, ε, για την υγεία και για την ε, δημόσια υγεία, συγκεκριμένα μελέτες από το 10 έως το 13, με στόχο να εντοπιστούν οι χημικές ουσίες ε, που εκπέμπονται από αυτά τα προϊόντα όπως είναι τα καθαριστικά, τα κοσμητικά χώρα, είδη προσωπικής ε, χώρου, είδη προσωπικής υγιεινής κτλ. Και να δούμε κατά πόσον υπήρχε κίνδυνος για τους καταναλωτές από αυτά τα προϊόντα. Τα επίπεδα έκθεσης μειώνονταν με, με, μία, με ένα προϊόν ε, σε μια περίπτωση. Επίσης, έχουν ε, κάνει μελέτες και ενώσεις καταναλωτών. Εκεί παρατηρούνται υψηλά επίπεδα παρόλα αυτά. Σε αρωματικά κεριά ή στα... ή τα αρωματικά στίκ που ανάβουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρουσία χημικών ουσιών, υπάρχει το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών, τα συστατικά, η τικετοθεσία. Σε ό,τι αφορά τη δε νομοθεσία, τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται στην ε, Γενική Οδηγία για Ασφάλεια των Προϊόντων, η οποία απαιτεί τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά να είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Αυτή είναι η υποχρέωση για τους ε, κατασκευαστές. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά να είναι ασφαλή και να μην περιλαμβάνουν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον καταναλωτή. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να το αποδείξουν την ασφάλεια στο προϊόν τους. Και αυτό μπορούν να το κάνουν ε, τηρώντας ε, τις προδιαγραφές που προβλέπει η Επιτροπή Επίση, η ΣΕΝ, ε, να τηρούν δηλαδή, τα σχετικά πρότυπα. Και υπάρχουν πρότυπα πράγματι, τα οποία έχει ορίσει η ΣΕΝ, ε, και αφορούν τα όρια πομπών, την πληροφόρηση του καταναλωτή και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα την συγκεκριμένη νομοθεσία για τα χημικά και για τα αποσμητικά, αυτά συνήθως είναι μείγματα χημικών ε, ουσιών, επομένως καλύπτονται από την νομοθεσία που λέγεται CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων. Υπάρχουν λοιπόν απαιτήσει για την ε, επισήμανση. Τι θα περιλαμβάνει η ετικήτα όταν ε, υπάρχουν κάποια χημικά ή αλλεργιογόνα συστατικά. Και ε, ο κανονισμό REACH εφαρμόζεται, ο οποίο επιτρέπει τον περιορισμό κάποιων χημικών ουσιών που θα μπορούσαν να είναι, έχουν υπάρξει αποδείξω ότι είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό. Από τον κανονισμό Ρίτς λοιπόν ήδη απαγορεύεται η χρήση μίας από αυτές τις χημικές ουσίες το 1,4 τρικολοβενθένιο και θα μπορούσαν οι περιορισμοί αυτοί να επεκταθούν να καλύψουν και άλλες ουσίες. Θέλω επίσης να πω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και για την επαγρύπτηση της αγοράς. Και όταν απαντούν τέτοια προϊόντα θα πρέπει να προβαίνουν σε κοινοποίηση μέσω του δικτύου γρήγορου, γρήγορης προειδοποίησης, το RAPEX. Το 2016 υπήρξαν 16 τέτοιες κοινοποίησεις για αποσμητικά, τα οποία εξέπεμπαν μία επικίνδυνη ουσία. Και πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην εκτίθεται καταναλωτέ σε επικίνδυνε χημικέ ουσίε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πράγματι οδηγία για την ε, ε γενική προστασία, το ΡΕΠΕΞ όπως είπατε και νομίζω ότι έχετε καλύψει διεξοδικά και εξαντλητικά. Θα φυσικά και οι συνάδελφοι μπορούν να ζητήσουν ε, το λόγο αν το επιθυμούν. Δεν βλέπω κανείς όμως να θέλει να λάβει το λόγο. Επομένως, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε, είδε τις διάφορες μεθόδους. Έχουμε και την οδηγία τη Γενική για την Ασφάλεια και το ΡΕΠΑΞ, το ε, σύστημα και προειδοποίησεις ε, για των προϊόντα και νομίζω ότι με αυτή την επικαιροποιημένη παρουσίαση μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά και να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η 1379 αναφορά για την προστασία ζώων και ανθρώπων από τα φυτοφάρμακα και τις τοξίνες. Είναι εδώ ο δόκτωρ Μέναχε. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gisela Ohr. Ε, γεια σας. Ε, λέγομαι Κιζέλα Ohr από την ε, Οργάνωση για την Προστασία των Ζώων και ε, στηρίζεται η αναφορά μου και από ε, τους συναδέλφους στους οποίους θα δώσω τώρα το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μου δίδεται να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπέβαλαν αυτήν την αναφορά και ο λόγος που την υποβάλαμε είναι ότι νιώθουμε ότι το REACH, ο κανονισμός REACH ε, υπό την παρούσα μορφή ε, δεν προστατεύει την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο λόγους. Ε, καταρχάς ότι βασίζεται σε δεδομένα από πειράματα σε ζώα και δεύτερον ότι δεν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα σχετικά με τις συνέπειες σε ανθρώπους. Ως κτηνίατρος ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ένα φάρμακο για άλογα δεν θα το ε, δοκιμάσω σε παπαγάλους. Γιατί λοιπόν ε, χρησιμοποιούμε ποντίκια ή αρουραίους για να δοκιμάσουμε φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπους. Ας μιλήσουμε για τη δυσπενόλη α. Τέθηκε στην αγορά μετά από δοκιμές σε ζώα. Ε, ο βιομηχανικός τομέας μπορεί να επιλέξει μόνος του ε, τα ζώα στα οποία θα κάνει τις δοκιμές ε, και το ε, συγκεκριμένο ποντίκι που, χρησιμοποιήθηκε ε, είναι κατά 100 φορές πιο ανθεκτικό στην δυσβενόλη α από ό,τι άλλα είδη ποντικιών και γι' αυτό ακριβώς αυτό το είδος επέλεξε η βιομηχανία για να ε, δοκιμάσει τη δυσφενόλη α. Η δυσφενόλη α είναι ενδοκρινικός διαταράκτης και όσοι γνωρίζετε πώς λειτουργούν αυτοί οι ουσίες γνωρίζουν ότι δεν είναι η ποσότητα που καθορίζει τις συνέπειες. Διότι για τη δυσφενόλη α, ελάχιστα μέρη ανά τρισεκατομμύριο ακούν για να κάνουν ζημιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσουν τις δοκιμές που γίνονται για την προστασία των ανθρώπων αλλά με βάση στοιχεία από δοκιμές σε ζώα. Δεύτερον, ο δεύτερος λόγος ε, που το REACH δεν προστατεύει επαρκώς ε, την υγεία των ε, πολιτών είναι ότι αγνοούμε τον μεγάλο όγκο ανθρωπίνων δεδομένων που δεν συλλέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και μιλώ για ανθρώπους από την αυτοκινητοβιομηχανία ή από οποιονδήποτε βιομηχανικό τομέα. Θα μπορούσαμε να λάβουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών από τους ανθρώπους αυτούς. Μόλις το Δεκέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα πρόγραμμα διοπαρακολούθησης ανθρώπων με βάση το ορίζον 2020. Πολύ αργά όμως. Διότι από το 2003 και μετά γνωρίζουμε ότι βρέφοι που γεννώνται έχουν ε, πολλά βιομηχανικά χημικά στο σώμα τους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά ουσιών, έχω έναν κατάλογο με 174 ε, ουσίες η εξέταση των οποίων θα έπρεπε να, ξεκινήσει το 2000, να είχε ξεκινήσει το 2007 με προτεραιότητα σε 300 χημικές ουσίες που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να μην σας συγκλονίζει ότι ε, η ε, πρωταρχική αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 14 ετών ε, στον δυτικό κόσμο σήμερα, η βασική αιτία θανάτου είναι ο καρκίνος. Εάν δεν σας συγκλονίζει αυτό, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σας συγκλονίσει. Από τη δεκαετία του 50 και του 60 γνωρίζουμε ότι ο καπνός ε, οδηγεί σε καρκίνο με βάση επιδημιολογικά δεδομένα. Ε, αν θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, θα πούμε ότι δεν ε, συλλέξαμε ανθρώπινα δεδομένα λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Εγώ όμως νομίζω ότι πρόκειται για εγκληματική αμέλεια. Το REACH μπορεί και πρέπει να προσαρμοστεί στην επιστήμη του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να σταματήσει η χρήση ζώων, διότι δεν μπορούν να, προβλε... να ε, προδικάσουν το τι γίνεται σε ανθρώπου, Ένα ποντίκι δεν ε, μπορεί να μα δώσει συμπεράσματα για αρουραίους. Όταν χρησιμοποιούμε τους κώδικες της Νιρεμβέργης του 47 και του 48, τότε έγινε νόμιμη η χρήση δοκιμών σε ζώα. Κυρίες και κύριοι, η νομοθεσία ε, βρίσκεται 70 χρόνια πίσω από την επιστήμη. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε την νομοθεσία, διότι οι δοκιμές σε ζώα δεν μπορούν να μας δείξουν τι γίνεται ε, με τους ανθρώπους. Έχουμε σήμερα τις σχετικές ε, τεχνολογίες, ε, έχουμε επιδημιολογία, έχουμε τιμωριακή επιδημιολογία, έχουμε διάφορες άλλες ε, τεχνολογίες. Ε, η τεχνολογία υπάρχει, η πολιτική βούληση χρειάζεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Απευθύνομαι στην κυρία Σούτετ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. να απαντήσω στους αναφέροντες ότι μέχρι ενός βαθμού συμφωνούμε. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι και εμείς θα θέλαμε ε, να βελτιώσουμε τις ε, επιστημονικές μεθόδους πρόγνωσης σε σχέση με τα πειράματα στα ζώα. Να τις βελτιώσουμε σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά θα πρέπει να σας πω κάποια σημαντικά σε σχέση με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει το έργο μας. Στο ΡΙΤΣ και σε άλλα νομοθετήματα όταν δεν υπάρχει εναλλακτική γίνονται πειράματα στα ζώα και ε, ε, αυτό ορίζεται από την οριζόντια οδηγία για την προστασία της χρήσης των ζώων και επιστημονικούς σκοπούς. Πρόσφατα, όπως λένε και οι αναφέροντες, για τα ζώα έχουμε το ΡΙΤΣ και την υπηρεσία την Ευρωπαϊκή ΕΚΑ έχει την έκθεσή της την τρίτη όσον αφορά την χρήση εναλλακτικών τεχνικών και όχι πειράματα στα ζώα για το ρίτσο. Με σε αυτή την έκθεση γνωρίζετε ότι τα βασικά δεδομένα προέρχονται από μελέτες ε, δοκιμών στα ζώα πριν τεθεί σε ισχύ το ρίτσο. Δεν έχουμε καινούργια δεδομένα από ζαό όμως για τα πιο περίπλοκα ζητήματα Γίνονται δοκιμές σε ζώα. Όπου ισχύει το ρίτς υπάρχουν κάποιες ε, ε, ενεργικές δυνατότητες που προτείνονται από την νομοθεσία. Και η χημική βιομηχανία χρησιμοποιεί την ε, σχάτη λύση που είναι τα ζώα. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τεχνολογική εναλλακτική. Τόσο αφορά τις μελέτες που έχουν γίνει για το ΡΙΤΣ μέχρι σήμερα. Έχουμε λιγότερα σπονδυλωτά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη μεριά έχουμε και λιγότερες πληροφορίες για τους διάφορους κινδύνους. Λιγότερους, λιγότερες πληροφορίες από ό,τι πριν αρχίσει να ισχύει το REACH η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη πασχίζουν τόσο ώστε σε τακτά διαστήματα να ενημερώνουν το ΡΙΤΣ όσον αφορά εναλλακτικέ. Όποτε αυτέ οι μέθοδοι μπορούν να μας δώσουν δόκιμα αποτελέσματα και επαρκή στοιχεία. Ε, αυτό γίνεται όσον αφορά τα σχετικά παρατήματα για δέρμα και μάτια. Αυτό αναφέρεται και από τους αναφέροντες. Η σχετική με τα πειράματα νομοθεσία ορίζει τι πρέπει να χρησιμοποιείται. 24 νέες μέθοδοι μέσα σε μια πενταετία έχουν ενημερώσει την νομοθεσία. Και πάνω από 70 ενημερώσεις συνολικές που θεσπίστηκε την νομοθεσία. Συμφωνούμε ότι το μέλλον της τοξικολογίας εξαρτάται από την κατανόηση των προβλημάτων. Οπότε οι νέες μέθοδοι θα πρέπει να στηρίζονται και σε κάποιες αρνητικές διαπιστώσεις. Πάντως, όλα αυτά που επεξεργάζεται τώρα μόνο ο ΩΣΑ και εμείς παρακολουθούμε. Δεν έχουμε κάποια διεθνή πρότυπα για το πώς ε, θα χρησιμοποιούνται νομίμως τα βρεθέντα εργαλεία. biomonitoring και διάφορες τεχνολογίες έχουν αναφερθεί από του αναφέροντες, σημαντικές τεχνολογίες. Όμως, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν αυτά τα εργαλεία να αντικαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα για τις πιο περίπλοκες ε, δοκιμές. Για την τοξικονομία προσπαθούμε να βρούμε κάποια ε, συμφωνία για το τι θα ισχύσει. Άρα χρειάζεται ακόμη χρόνο. Πριν μπορούμε αποδεκτέ και κάτω και από τον νόμο λύσεις. Υπάρχουν δυνατότητες όμως ακόμα και επομένως η διεθνείς κοινότητα προσπαθεί. Και όσα έχει συγκροτήσει κάποιε ομάδε εργασία, το ώστε μέχρι το, τα του 2018 να ε, έχει κάποιες καρπούς για τοξικονομία, για μεταβολισμούς, για, για διάφορους κλάδους της τοξικολογίας. Έχουμε από τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο. Έχουμε όμως και ευελιξία σε σχέση με το Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που δεν προέρχονται από πειράματα στα ζώα. Αλλού δεν υπάρχει τέτοια ευελιξία. Biomonitoring που μας δίνει κάποια δεδομένα που εάν είναι ισχυρά και βάσιμα επιστημονικά μπορεί να ληφθούν υπόψη. Κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αξιολόγηση ε, των πειραμάτων σε σχέση με το πόσο προστατεύει άνθρωπο και περιβάλλον και αυτό έγινε στην έκθεση αξιολόγησης του 2017. Πρόκειται να εγκριθεί ο κανονισμός αρχάς του 2018, οπότε στην έκθεση αυτή πρόκειται να αναλύσουμε τι συμβαίνει, πώς μπορεί να έχουμε περισσότερη ασφάλεια και συμφωνούμε ότι η συστηματική υλοποίηση της αρχής προφύλαξης στις διαδικασίες του REACH είναι κάτι που προϋποθέτει και περιορισμούς, απαγορεύσεις και αξιολόγηση. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξεργαζόμαστε όσο γίνεται πιο ε, προηγμένες τεχνολογίες και ευελιξία στην ε, ε, λήψη αποφάσεων, να υπάρχει προβληψιμότητα και τελικά να μειώσουμε τη χρήση των ζώων στα πειράματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουν το λόγο η κυρία Εύη πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αφετηρία μας είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο συρρυκνώνει τον προπολογισμό που καλύπτει την έρευνα των εναλλακτικών μεθόδων. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός. Κάθε χρόνο η περικοπή είναι γεγονός. Πρώτον αυτό. Δεύτερο γεγονός sperimentazione eh, Αυτό αφορά και το ότι ακόμη δεν έχουμε συγκρισιμότητα μεταξύ πειραμάτων σε ζώα και εναλλακτικών. Άρα χρειάζεται να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση. Συγκριτική. Τέτοια πειράματα να γίνουν όσον αφορά την έγκριση φαρμάκων και χημικών. Το λέει η ίδια η Επιτροπή. Παγίως. Ότι θέλει στο μέλλον, κάποια στιγμή που δεν την διευκρινίζει, να σταματήσουν τα πειράματα σε ζώα. Συμφωνώ 100% εγώ με την ε, αναφορά αυτή. Χιλιάδες την έχουν προσυπογράψει. Και αυτή αποτελεί ακόμα μία αναφορά. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες αναφορές και πολλές από αυτές κλείσανε. Και κλείσανε με πάρα πολύ επιφανειακή εξέταση, στο γόνατο. Και πάντοτε η Επιτροπή λέει για το ΡΙΤΣ, λέει για πρωτοβουλίες copy-paste κάνει για την ε, απάντηση στην ε, πρωτοβουλία των πολιτών, το ΙΤΣΕ. Ωραία για περισσότερο και αυτό τους ε, Ευρωπαίους και το ότι τέτοιου είδους εμβαλωματικές απαντήσεις δεν τους αρκούν. Ακόμα απομένουν πάρα πολλά πρέπει να γίνουν και σε πολιτικό επίπεδο. Συλλογή δεδομένων, ευαισθητοποίηση. Και όπως έλεγα υπάρχουμε εδώ αυτή την παρουσίαση των δεδομένων. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο δεν έχουμε είναι την πολιτική βούληση για ανάληψη δράσης. Επαναλαμβάνω. Να είναι ανοιχτή αναφορά. και η Επιτροπή μας να ξανασυζητήσει με τους αναφέροντες και να μην κλείνει τις σχετικές αναφορές. Και να μας πει επομένως δύο λόγια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συρρήγνωση του προπολισμού για τις αναλλακτικές και γιατί παγώνει οποιαδήποτε προσπάθεια ε, που έχει σχέση με την εγκατάλειψη των πειραματών στα ζώα. Ο πρόεδρος, έτερος. Then I'm happy to give the floor. Αν όχι να δώσω ξανά το λόγο στους αναφέροντες για δύο λεπτά. Αν επιθυμούν το λόγο βέβαια. Παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και η απόφαση να είναι υπέρ μας. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, μάλλον αν δεν συμβεί αυτό θα θέλαμε εγγράφος να ενημερωθούμε για να καταθέσουμε καταγγελία προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. I didn't, could Δεν σας ε, πολύ κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το πείτε λίγο με περισσότερα λόγια. Λέτε να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και τι άλλο λέτε. Εξηγήστε μας λίγο ποια ήταν η πρόθεση, τι εννοούσατε με αυτά που είπατε. Ich möchte, dass die Petition... Θα θέλαμε η αναφορά να ε, θεω... κλείσει θετικά για εμάς, δηλαδή να έχει θετική έκβαση, να παραμείνει ανοιχτή για να συζητηθεί εκ νέου και η απόφαση να είναι υπέρ μας. The point that I didn't Ναι, αυτό που δεν κατάλαβα ήταν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλετε εσείς, λέει η αναφέρουσα. You were mentioning in your... Η πρόεδρος, ε, Είπαμε, αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι αν κλείσει η αναφορά και δεν υπάρξει υπέρ μας απόφαση, θέλουμε εγγράφως να ε, μας το γνωστοποιήσετε για να καταθέσουμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι η υγεία και η προστασία της υγείας των ε, συμπατριωτών, των συμπολιτών μας. Τώρα αυτή τη φορά έγινε κατανοητή πρόεδρος μάλιστα. Δηλαδή λέτε είτε να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, αυτό ζητείτε, ή θα πάτε την Επιτροπή μας στο δικαστήριο. Μα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. like Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο όσο καιρό είμαι πρόεδρος. Της Επιτροπής Αναφορών και θέλω να σας πω ότι σε αυτήν την επιτροπή έχουμε μία συνάντηση, είχαμε μάλλον μια συναντηση ειχαμε μάλιστα μια το Σεπτέμβριο του 2016, όπου είχαμε αποφασίσει να επαναξιολογήσουμε και να συζητήσουμε τις αναφορές για τη γλυφοσάτη, που είναι μία από τις επιβλαβείς ουσίες μέσα σε 18 μήνες. Αυτό θα γίνει έξι μήνες από τώρα και θα πρότεινα ε, επομένως να παραμείνει ανοιχτή αναφορά όπως και κάποιες άλλες ε, αναφορές που έχουν το ίδιο θέμα και σε έξι μήνες από τώρα να τις ξανασυζητήσουμε και στο μεταξύ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Is that colleagues what we can do? Συμφωνείτε αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται νεύουν, συγκα... Συγκατα... οι συνάδελφοι, οπότε αυτή τη φορά γλιτώσαμε το δικαστήριο από ό,τι φαίνεται. Καλό είναι αυτό, κυρία Εύη. Madam Chair, can we also forward the petition to the Να διαβιβάσουμε και στην Επιτροπή ή κυρία Πρόεδρε, την αναφορά. Γιατί έχουμε στους επόμενους μήνες και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη χρήση ζώων σε εργαστηριακές δοκιμές. Θα ήταν καλό, ίσως έτσι θα επιταχυνόταν η συζήτηση και θα συμμετείχαν και οι πολίτες στην αναθεώρηση αυτή. Εξαιρετική πρόταση και πράγματι θα ενημερώσουμε και την Επιτροπή Ένβη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλό ταξίδι στους αναφέροντες. Και περνάμε στην επόμενη δέσμη αναφορών, το 22 θέμα δηλαδή τη μερικής διάταξη. έχουμε την αναφορά 130, την αναφορά 131, 134, 154 και 155. Είναι εδώ οι αναφέροντες, ένας για κάθε ένα από τα Κανάρια νησιά. Για την Τενερίφη λοιπόν έχουμε το Σαντιάγο Πέρεθα Γκαρθία. Ο κύριος Μάτο, διαδικαστικό, παρακαλώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μάτο, ναι, ένα ερώτημα. Ένα διαδικαστικό μάλλον, κυρία Πρόεδρε. Αν είχα καταλάβει καλά, οι εν λόγω αναφορές θα έμπαινα στη μέση διάταξη, αλλά αν είχαμε λάβει τις ε, εκθέσεις της Επιτροπής και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα και χαίρομαι που είναι εδώ οι αναφέροντες, τους προσκαλέσαμε, ήρθαν εδώ και είπα ότι θα συμπεριφερθώ καλά και αυτό και θα κάνω. Δεν έχω πρόβλημα και καλά κάναν και ήρθαν οι άνθρωποι. Αλλά σας παρακαλώ ή να μην βάζουμε στην μερσιά διάταξη ε, τέτοια ζητήματα αν δεν έχουμε ε, τις εκθέσεις, τις σχετικές, τα σχετικά έγγραφα ε, ή εντάξει, να τους καλούμε όταν έχουμε στη θέση μα όλα τα έγγραφα. Όχι ότι έχω πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση που ήρθαν οι άνθρωποι εδώ. Παναλαμβάνω. Η πρόεδρο. Ακούστε, είναι σήμερα αυτές οι αναφορές ε, μετά από την απόφαση που έλαβαν οι συντονιστές στις 10 Ιουλίου. Τότε αποφάσισαν οι συντονιστές, πλειοψηφία τους, τα θέματα αυτά να συμπεριληφθούν στη σημερινή μερίσια διάταξη. Και γι' αυτό τώρα με χαρά μπορώ να κηρύξω την άνοιξη της συζήτησης για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τις αναφορές αυτές και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Σαντιάγο Πέρεφ, Γκαρθία για την 130 αναφορά. Νομίζω έχετε να μας δείξετε και ένα PowerPoint. Okay, so here we go. And... Ξεκινάμε λοιπόν, Τενερίφη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές. Εάν νόμος κράτος μέλους ή άλλες οντότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει την άδεια σε κάποιο δημόσιο φορέα να αυτοεξαιρείται από την ε, ένομη τάξη, τότε δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση να προβαίνει σε απαλατριώσεις με κάποιο είδους ε, αποφάσεις που φέρνουν δυσμένες διακρίσεις τα οι οποίες εκφεύγουν της χωροταξίας. Γιατί έχουμε τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχει η διάκριση εξουσιών και αυτό όσον αφορά την έγκριση κάποιων προγραμμάτων και σχεδίων για το περιβάλλον. Οπότε έχουμε μια συνταγματική τάξη που δεν επιτρέπει στους τακτικούς δικαστές το, την, αναστολή εφαρμογή ε, του νόμου και έχουμε επομένως νομοθετήματα της διοίκηση που έχουν βέβαια την, το, το, το εκμύριο της νομιμότητος αλλά υπάρχει επίσης και το θέμα της συνθήκης του άρχους και του θεμελιώδους δικαιώματος ε, της, του δικαστικού ελέγχου όπως το άρθρο 47 αυτής της συμφωνίας. Θέλουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν, υπάρχει το δικαίωμα στην ισότητα, στην ε, ιδιοκτησία, το προστασία του περιβάλλοντος και στην δικαστική προστασία. Και επίσης πρέπει να υπάρχουν οι βασικοί μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκαιο κατησχύει σε αυτή την περίπτωση. Πρόκειται τώρα για κάποια απειλή κατά του περιβάλλοντος και κατά των φυσικών πόρων των Καναρίων. Και με νόμο αυτά κατοχυρώνονται, δηλαδή η προστασία αυτού του περιβάλλοντος όσον αφορά τον νόμο για τη γη και την προστατευμένους χώρους τέλος πάντων. Και τώρα ε, Υπάρχουν αυτό το νόμο που ψηφίστηκε με μεγάλη συνένεση. Υπάρχουν κάποια όρια στην ανάπτυξη. Αυτός ο νόμος για τη γη ε, έχει σκοπούς ε, απλούστευσης και απορρίθμισης αλλά ουσιαστικά είναι κατά της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωθεί στη χρήση φυσικών πηγών που δεν είναι, φυσικών που δεν είναι ανανεώσιμη. Αυτού του είδους ο νόμος αφορεί, αφορά την χωροταξία των Καναρίων και εδώ υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες διατάξεις. Και ο κοινό σε αυτών των μέτρων αυτού του νόμου είναι ότι αλλάζουν οι κανόνες του σχεδιασμού ε, για το περιβάλλον πέραν των όσων διαδικασιών προβλέπονται. Παρά την σχετική του 2003-35 αυτά είναι τα σχέδια ε, ενδιαφέροντος ε, νησιωτικού ή της αυτόνομης διοικητικής περιφέρειας. Και έχουν να κάνουν σχέση με τον τουρισμό, τα πολιτιστικά, τη βιομηχανία, τον αθλητισμό και λέει αυτός ο νόμος ότι είναι δυνατόν αυτόνομα να ληφθούν μέτρα για όλους αυτούς τους ε, τομείς. Οπότε μπορούν να διακηρύξουν κάποιο μέτρο ότι είναι ε, για το δημόσιο κοινό καλό ή για το κοινωνικό ενδιαφέρον. Και έχει κάποια αφιολογήματα μέσα αυτός ο νόμος και χρησιμοποιεί κάποιες διατάξεις για να εννοήσει κατά παρέκκληση της κείμενης νομοθεσίας. Όμως έτσι δεν έχουμε χώρο ταξία, δεν έχουμε έτσι σχεδιασμό. Είναι κάποιο είδους σχέδια εκτελεστικά, ούτως ώστε να εξαιρεθούν αυτά τα σχέδια από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δυναμητίζονται θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει εγγύσεις. Το σύστημα του κοινωτικού δικαίου αφορά τον, στο χώρο και χρόνο την υλοποίηση κάποιων αξιών. Και αυτός ο νόμος για τη γη εμποδίζει την πρόσβαση στους πολίτες στην ε, νομοθεσία για τα θέματα τα περιβαλλοντικά παρά την συνθήκη του άρχους. Παραβιάζει την ισότητα και έτσι ματιώνει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Επομένως έχουμε τώρα καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατηγορώνεται από τον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και όλα αυτά αντιβαίνουν σε οδηγίες, σε διάφορα νομοθετήματα Έχουμε το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 191 τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. Επίσης ε, έτσι παραβιάζονται και οι Ισπανικοί νόμοι μεταφοράς. Για 3-4 δεν σας το λόγο διακόπτει ο Πρόεδρος. Τώρα τον έχετε υπερβεί κατά 100%. Τι θα γίνει και οι φίλοι, οι συνάδελφοι από τα άλλα νησιά δεν θα πρέπει και αυτοί να λάβουν το χρόνο. Παρακαλώ, προσπαθήστε τώρα να κλείσετε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να μείνει ανοιχτή η αναφορά και το Κοινοβούλιο να ασκήσει τον έλεγχό του και μέσω της Κομισιόν να πιεστεί η κυβέρνηση της χώρας μας ούτως ώστε να ισχύσει όπως προβλέπεται το κοινοτικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα από την Λαπάλμα έχουμε την Βανέσα Καταλάν Γκονσάλες. Τρία με τέσσερα λεπτά το πολύ λέει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι από τη Λαπάλμα. Ε, έχουμε 700 τετραγωνικά και το, η UNESCO την θεωρεί προστατευόμενη περιοχή. Έχει μεγάλη συγκέντρωση, μεγάλη βιοπικιλότητα, πάνω από 490 ή 240 μόνο στη Λαπάλμα απαντούν. Το μισό, ε, η μισή επιφάνεια της ξηράς και το 1 τρίτο των υδάτων είναι προστατευόμενα από την UNESCO. Υπάρχει όμως ε, η απειλή από αυτό το νομοσχέδιο, γιατί μπορεί να επιτρέπει την ε, άναρχη δόμηση και να καταργηθούν τα φυσικά εδάφη που και να πληγεί η πολιτιστική κληρονομιά, το τοπίο, ε, το περιβάλλον. Και μιλάμε για περιοχές που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε πολεοδομικό ιδιωτικό ή δημόσιο σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εδαφική χωροταξία και τα σχέδια. Με αυτό το νομοσχέδιο όμως θα εφαρμοστούν σχέδια δόμησης που προέρχονται από τα προγράμματα πολεοδομίας ε, τουριστικής ανάπτυξης ε, που έχουν ε, ακυρωθεί από το δικαστήριο. Πρέπει να γίνει λοιπόν στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Είναι μια υποχρέωση από την Οδηγία 42 του 2001. Επίση, πολλά από αυτά τα προγράμματα που έχουν ακυρωθεί και θα τα σώσει αυτός ο νόμος, επαναλαμβάνω δόμηση ή ένα γήπεδο γκόλφα, έχουν να κάνουν με δίκτυα περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και έχουμε κατά την οδηγία 43 που έχει να κάνει με την διατήρηση των οικοσυστημάτων, την χλωρίδα και την πανίδα. Βλέπετε εδώ στην Ταμάνκα έχουμε μια προστατευόμενη περιοχή γεωλογικοί σχηματισμοί, ηφαιστειακοί σχηματισμοί, λάβα και ενδυμικά είδη ε, χλωρίδας και πανίδας που ορισμένα εντάσσονται στα απειλούμενα είδη, στα είδη ύπος ε, προστασία. Υπάρχει κίνδυνος ε, και για διάφορα είδη που τα βλέπετε εκεί. Ζητούμε να μην επιτρέψετε την καταστροφή του τοπίου, της φυσικής κληρονομιάς μας που είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο προσεκύουμε τους ε, τουρίστες. Να μην καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε στην περιοχή μας και να προστατεύουμε την κληρονομιά μας. Thank you very much. And a master... Σας ευχαριστώ πολύ. Είδατε πόσες πληροφορίες... μπορέσατε να συσσωρεύσετε, να στριμώξετε όλες αυτές τις ε, πληροφορίες σε μια τόσο γρήγορη σύντομη παρουσίαση. Ε, ο κύριος Μαρτίνεφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Κάλλης. Πέρασε όλες και όλους. Προέρχομαι από την Γομέρα. Εδώ έχουμε ποικιλία στο περιβάλλον, 470 ε, χιλιόμετρα και έχουμε 4.082 είδη στη γη και 1021 είναι από τα Κανάρια και 224. Βλέπετε ότι έχουμε την περισσότερη ενδημία στην Ευρώπη ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και 25 ζώνες έχουμε το φυσικό πάρκο του Χονάι και αυτό αποτελεί με τις παγκόσμιες κληρονομιάς και εκεί πέρα έχουμε επίσης ένα οικοσύστημα στον αφορά το τοϊκή ε, δάσος και αυτό έγινε στην τριτογενή περίοδο, δημιουργήθηκε τότε που από την Ευρώπη αυτά τα είδη εξαφανίστηκαν. Το 2008 είπαμε ότι έχουμε ε, την Ευρωπαϊκή Κάρτα του Βιώσιμου Τουρισμού και τότε είπαμε ότι όλα τα οι φυσικοί χώροι ε, εκπροσωπούνται και καλύπτονται και έχουμε ε, τώρα μια βιώσιμη ανάπτυξη για έναν τουρισμό εκεί που προστατεύονται αυτά τα εδάφη και όλα αυτά η UNESCO τα θεώρησε ως προστατευμένο χώρο για την παγκόσμια βιοσφαίρα. Οπότε έχουμε τα καινούργια σχέδια για έναν τουρισμό στην Πάλμα και αυτό ε, αφορά την αναφορά που τώρα σας υποβάλαμε και ε, τίθενται να αμφιβόλο όλα αυτά τα μέτρα ε, προστασίας που είπαμε. Και έτσι δεν υπάρχει βιώσιμος τουρισμός. Δεν υπάρχουν εγγύσεις για βιώσιμη διακήρυξη είναι κατά του πλαισίου δράσης ε, για μια διαχείριση βιώσιμη και δεν υπάρχει κάποιο είδους χωροταξία και των, και των νόμων για τη χρήση της γης. Και επίσης δεν υπάρχει κάποιο είδους ολοκληρωμένη αντίληψη και ε, σφαιρική και βάζει την γεωργία στο περιθώριο δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ούτε ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται και σε καμία στιγμή, σε καμία φάση της νομοθεσίας αυτής δεν προβλέπεται κάλυψη όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων. Δεν ε, λαμβάνεται όψη αρχή της προφύλαξης, δεν υπάρχουν ε, κάποιο είδους ε, όρια των παρεκκλήσεων για την ανάπτυξη. Ε, από όλους μας εξαρτάται ένα τέτοιο νησί να μπορεί να διασωθεί και να προστατευτεί με όλες του τις ιδιομορφίες. Ιέρο. Χουάν Ραμόν Γκονθάλεφ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Εγώ έρχομαι από την ε, ε, Ιέρο, αυτό την Ίσο των Καναρίων και ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τους ευρωβουλευτές. Ο στόχος της παρουσίασής μας είναι να καταγγείλουμε το νόμο των πράσινων νησιών, πολύ μεγάλος εφημισμός. Ήρθα εδώ γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βλάψει σοβαρά και ανεπανόρθωτα την συνίσωση Ιέρο, Γκομέρα και Λαπάλμα αυτό ο νόμος, γιατί άλλωστε καταπατά και το περιβαλλοντικό δίκαιο. Έχουμε 268 τετραγωνικά χιλιόμετρα και λίγο πάνω από 10.000 ε, κατοίκους με βάση τα επίσημα στοιχεία. Τα Κανάρια νησιά είναι άκρο από κέντρο περιφέρεια και η πιο απομακρυσμένη είναι, η νήσος ελιέρο. Δεν υπάρχει επαρκή σε θαλάσσια και ενέργεια ε, διασύνδεση για να αναπτυχθεί η οικονομία. Υπάρχουν επίσης ε, τα μέσα τουριστικής, ε, τουριστικού σχεδιασμού και έχουν λάβει χώρα μια σειρά από ε, project ε, δυνάμει αυτού του νόμου τα οποία θα επηρεάσουν ε, το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τη χλωρίδα και Πανίδα. Το Ιέρο έχει σημαντική πολιτιστική φυσική κληρονομιά, κυρίως είναι πλούσιο σε συγκεκριμένα είδη ζώων και φυτών, όπως παραδείγματο χάρη γιγαντέα σάβρα του Ελιέρο και 11 είδη ενδυμικής πανίδας. Η UNESCO θεωρεί ότι είναι ε, προστατευόμενος χώρος της βιοσφαίρας ε, το 2000 και το Χέο Πάρκε το 2014. Ε, είναι ένα γεωλογική κληρονομιά. Καλύπτει το σύνολο του νησιού Είναι ένα φυστογενέ νησί το Ιέρο και αυτό το ε, βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα σε αυτό το γεωλογικό πάρκο. Το 60% ε, του εδάφους του Ιελιέρο προστατεύεται. Είναι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 ε, ή στο Δίκτυο των Καναρίων. Είναι φυσικό μνημείο, έχει προστατευόμενα τοπία, διάφορα άλλα εθνικά πάρκα κτλ. Θέλω να τονίσω το φυσικό πάρκο της Φροντέρα S702041 που είναι μια ειδική ζώνη διατήρησης και που θα επηρεαστεί πολύ περισσότερο με αυτό το νόμο. Έχει 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή ε, ετοιμάζεται ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο ε, στο νότο του Ελιέρο και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες συντήρησης, να γίνουν επιστημονικές σπουδέ και να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο το νησί. Θα πρέπει να φροντίσουμε τη φύση, όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη. Δεν πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών και της φύσης. Πρέπει να προχωρήσουμε σίγουρα αναπτύσσοντας ε, το νησί οικονομικά αλλά με οικονομική και κοινωνική αηφορία να προασπίσουμε το φυσικό μας περιβάλλον στο οποίο μέσα ζούμε. I thank you very much and extend immediately. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να δώσουμε τη συνέχεια της κοιτάλης στον Αντώνιο Πέρεθ, ο οποίος προέρχεται από την Γκραν Κανάρια. <clears throat> Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Εδώ βρισκόμαστε κυρίως γιατί το αρχιπέλαγος των ε, Καναρίων είναι μοναδική βιολογική περίπτωση στον κόσμο. Μιλούμε για 7.747 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 22.000 ε, είδη, από τα οποία 3.700 είναι ενδυμικά ε, και ζουν στα δάση. Έχουμε 220 ζώνες που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Πρόκειται για μια, έναν φυσικό πλούτο και πλούτο του περιβάλλοντος και μαζί με το κλίμα, την οικονομική ανάπτυξη ε, έχουμε μια τουριστική δραστηριότητα και φτάσαμε τα 15 εκατομμύρια επισκεπτών και έγινε μια έκρηξη δημογραφική και τουριστική δεκαετία του 60 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Όμως ε, η χωροταξική αναρχία έπληξε το περιβάλλον. Η πνευματική ισορροπία διατεράχθη. Στη δεκαετία του 90 και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα περάσανε κάποια νομοθετήματα στο περιβάλλον που ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλε τις πτέρυγες και ακολουθήσαμε τον ΟΗΕ, το Συμβουλίο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητά μα τα όσα επιτάσσει η προστασία του κοινού μέλλοντος, αλλά και οι συνθήκες ε, ή διεθνεί για το περιβάλλον. Στο αρχιπέλαγος αυτό τώρα βρισκόμαστε στα όρια μας όσον αφορά ε, τον φόρτο ούτως υπήν. Αυτό φαίνεται από το οικολογικό αποτύπωμα, όπως ήδη έχει υπολογιστεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ε, πυκνότητα ε, όσον αφορά τη, τον κόσμο και τους τουρίστες. Οπότε ο στόχος μας τώρα είναι να έχουμε ένα τουριστικό μοντέλο που να είναι ένα πρότυπο ποιότητας όπως θέλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μιλάμε για το 25% ε, στον τομέα που έχουν πέσει σε ανεργία, στον τομέα των τουριστικό. Έχουμε σχετικές, ε, σχετικά νομοσχέδια το 2017 που προσπαθούμε να καλύψουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Αυτός ο τουρισμός all inclusive δεν έχει σχέση με το ποιοτικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το επιθετικό αλλά αυξάνεται. Οπότε τώρα έχουμε αυτή, αυτή τη νέα χωροταξική νομοθεσία κατά τη γνώμη μας. Η νέα νομοθεσία όμως αντιβαίνει στην ισορροπία που υπήρχε μεταξύ βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Τώρα περνάνε κάποιοι νόμοι με απλή πλειοψηφία. Ας μην μιλήσουμε για το εκλογικό μας σύστημα. Γιατί οι εκπρόσωποι αυτών των πλειοψηφιών ε, ε, συγκεντρώνουν λιγότερες ψήφου λόγω του συστήματο από αυτού που ψηφίζουν κατά αυτών των νέων νομοθεσιών. Θέλουν κάποιο είδου γρήγορη και αχαλήνοτη ανάπτυξη και να μην υπάρχει ούτε έργο, ούτε χωροταξία, ούτε τίποτα. Και θα πρέπει επομένω να δούμε το πώ θα υπάρξει κοινωνικό και κρατικό έλεγχο. Θα χρειάζεται να ισχύσει η αρχή τη προφύλαξη, ε, να κατησχύσει παντού για κάθε είδου πανέβαση στο χώρο στο περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει από την αυτόνομη διοίκηση. Διακόπτει ο προέδρο. Κοιτάξτε, μας πιέζει ο χρόνο θα πρέπει να κλείσετε, γιατί οι περισσότεροι ξέρουν τον περιεχόμενο των αναφορών. Α, μάλιστα λέει. Επομένω με λίγα λόγια νομίζουμε ότι αυτή η νομοθεσία η οποία τώρα θεσπίζεται στην αυτόνομη δική μας περιφέρεια ε, προσπαθήνουμε με επίγοντα τρόπο να ε, βγάλει τους πολίτες από τη διαδικασία της χωροταξίας και σχεδιασμού του περιβάλλοντος. Και από τον είναι τέλος την κατάσταση. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ και εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Καναρίων, Κριστίνα Ντελεόν Παρέρο. Σας καλώ να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση των Καναρίων ευχαριστεί ιδιαίτερα στην πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών και τους ε, λοιπούς ευρωβουλευτές που τη έδωσαν τη δυνατότητα να εκθέσει την άποψή τη. Ε, και θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι αλλά περιμένω να δείξετε την ε, γενοδορία σας και εσείς, γιατί πρέπει να αναφέρουμε πέντε διαφορετικές αναφορές. Η μία αναφορά τον ε, νόμο για, το, για τη χρήση του εδάφους, οι τέσσερις αφορούν άλλο νόμο, τον νόμο που λέγεται νόμος ε, των πράσινων νησιών και αφορά ουσιαστικά την τουριστική δραστηριότητα Γομέρα, Ελιέρο και Λαπάλμα. Εγώ έχω γεννηθεί στην ε, Τενερίφη, ζω στην ε, Γκραν Κανάρια και ε, ο άντρας μου έρχεται από τη Λαπάλμα, που σημαίνει ότι εκπροσωπώ ουσιαστικά σχεδόν όλα τα Κανάρια νησιά. Βέβαια, αυτό το οποίο όλους μας μας ενδιαφέρει ως Κανάριος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Τα Κανάρια όπως είπαν και οι αναφέροντες, είναι ένα αρχιπέλαγος από έχει 7 νησιά και εξαιρετικό φυσικό πλούτο. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο το έδαφος ε, την χάνει περιβαλλοντικής προστασίας ε, κατά το 50% της εκτασής του. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή σημασία στην αυστηρή συμμόρφωση της περιβαλλοντικής και εδαφικής νομοθεσίας. Η εδαφική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την Ισπανία γενικά, το βασίλειο της Ισπανίας, είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, των αυτονομιών. Γι' αυτό στα εδαφικά ζητήματα έχουμε πλήρη αρμοδιότητα εμείς κυβέρνηση των Καναρίων. Όπως είπα, έχετε πέντε καταγγελίες, πέντε αναφορές λάβει. Οι τέσσερις αφορούν τον νόμο που ε, επηρεάζει, που αφορά μόνο τα νησιά Ελιέρο, Λαπάλμα, Λαγομέρα. Και υπάρχει και μία αναφορά που αφορά έναν πρόσφατο νόμο, τον νόμο για το έδαφος, για τη γη. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο νόμο, Ένα εκπρόσωπο από κάθε νησί μίλησε για αυτόν τον νόμο. Ο πρώτο νόμο λοιπόν προτείνει ένα μοντέλο τουριστική ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμο και θα αφορά ειδικά το κάθε νησί. Ακριβώ επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το οικοσύστημά του, που βασίζεται ουσιαστικά στην διατήρηση των φυσικών πόρων με την ε, προώθηση τουριστικών εγκαταστάσεων μικρών διαστάσεων ή μεσαίων διαστάσεων για να υπάρχει μια συντηρητική ανάπτυξη για να μην υπάρξει αυτή η απερίμωση που βλέπουμε σε, αυτό το, σε αυτά τα μικρά νησιά. Ενώ αντίθετα ε, στα ε, πιο τουριστικά δραστηριοποιούμενα νησιά υπάρχει υπερπληθυσμός και δεν το κάνει αυτό μόνο ο κυβέρνηση των Καναρίων. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, ε, κάντε και αυτό που έκανα ε, που προετοιμάζοντας την παρέμβασή μου έψαξα στο ίντερνετ βάζοντας ε, στη μηχανή αναζήτησης το νόμο για τα πράσινα νησιά ή το, ρόλο, το νόμο 2 του 2016 που τότε γκρίφτηκε δηλαδή το 2016 και βρήκα πάρα πολλά σχόλια ένα θα σας πω μόνο η Δόνια Εύα Μπλάνκο εδώ που είναι υπεύθυνη για τη μονάδα έρευνας και κατάρτισης του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Περιβαλλοντικού Δικαίου η οποία λέει ότι αυτός ο νόμος είναι παράδειγμα, καλό παράδειγμα προτάσεων τον εξορθολογισμών των τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά αυτά. Κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα υπόδειγμα, ε, είναι ένα μοντέλο για την, ε, το συμψηφισμό μεταξύ οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης και μιας βιώσιμης ανάπτυξης περιβαλλοντικά που σέβεται το περιβάλλον και αποτρέπει την απερίμωση. Πέραν και σε αντίθεση με αυτά που θέλησαν να πούν ή είπαν τελικά οι αναφέροντες, συγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2016 με 80% των ψήφων ψήφων ψήφισαν όλα τα μεγάλα κόμματα υπέρ. Και το φιλελεύθερη, και το λαϊκό και το σοσιαλιστικό κόμμα ψήφισαν υπέρ. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τον νόμο των τριών αυτών νησιών, Ιέρο, Μέρα, Πάλμα. Όλοι οι βουλευτές που εκπροσωπούσαν αυτά τα τρία νησιά, τα πράσινα νησιά όπω τα λέμε και όλοι στο σύνολό του ανεξαρτήτω πολιτικής ε, τοποθέτησης ψήφισαν υπέρ. Κάτι ακόμη πιο σημαντικό, όλε οι κυβερνήσει ε, των ε, εταιριών αυτών νησιών συμφωνούσαν και είχαν κάνει πρόταση υπέρ αυτού του βιώσιμου μοντέλου. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό αν θέλετε, οι Δήμοι των νησιών αυτών είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτό το μοντέλο βιώσιμη ανάπτυξη. Ο νόμο σέβεται πλήρω την περιβαλλοντική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία, θα υπήρχε μεγάλο κίνδυνο ε, για τα νησιά αυτά που βασίζονται στην προσέγγιση φυσική κληρονομιά. Δεν θέλω να σας, ε, να σας παρακουράσω με νομικά ζητήματα. Μπορείτε να διαβάσετε τον νόμο και μπορείτε να δείτε κάθε ένα από του νόμου και θα δείτε ότι όλα αυτά τα μέσα χωροταξίας που προβλέπει ο νόμος δημιουργούν μετά μια διαδικασία με περιβαλλοντική ανάλυση, περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με την οδηγία. Υπάρχει δε πλήρη συμμετοχή των πολιτών, δημόσια ενημέρωση. Δημοσιεύονται δε στις εφημερίδες με το μεγαλύτερο τυράζ όλα αυτά και δίνονται απαντήσει στου ισχυρισμού και στι καταγγελίε. Αν δεν υπήρχε αυτό ο νόμο, όπω είπα, υπήρχε μεγάλο κίνδυνο για αυτό το μοντέλο που δημιουργείται ε, από τα νησιά αυτά, που βασίζεται η βεβαίωσή του στην προστασία τη φυσική κληρονομιά. Με τον νόμο αυτό, η πρόεδρο, θα μπορούσατε να συνοψίσετε, έχετε ξεπεράσει ήδη τα πέντε λεπτά που είχατε στη θέση σα. Ευχαριστώ. Τρία δευτερόλεπτα αν μου επιτρέπετε, μόνο για να πω δύο πράγματα. Και μόνο για ένα θέμα μίλησα, για τον νόμο για τα πράσινα νησιά. Έχουμε και τον νόμο για τη γη, για το έδαφος. Πούτε και αυτή η νομοθεσία καταπατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα γίνει η περιβαλλοντική αξιολόγηση και θα συμμετάσχουν, θα ενημερωθούν και οι πολίτες. Το Συνταγματικό Δικαστήριο ε, και τα άλλα αρμόδια όργανα έχουν ε, την αρμοδιότητα ε, και την δικαιοδοσία. Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το συνταγματικό δικαστήριο θα, το, θα ε, του ζητήματος. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα. Στόχος μας είναι να τηρήσουμε αυστηρά την ε, βασική σπανική νομοθεσία αλλά και την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να κλείσουν οι αναφορές γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Και αν μείνουν ανοιχτέ αυτό δεν θα στηρίζεται ούτε στο δικαίωμα της συμμετοχής των πολιτών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Ντάνιελ Φερνάντες Κόμες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους ε, αναφέροντες και την ε, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διοίκησης για τα όσα μας εξήγησαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει γνώση κάποιων από τα στοιχεία που εδώ εκτέθησαν μέσω των καταγγελιών που έχουν γίνει. Έχουμε λάβει τα στοιχεία και τα έγγραφα στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος πρόσφατα. Όμως ακόμα δεν είχαμε βρει το χρόνο να μελετήσουμε εις βάθος όλο αυτό το υλικό και ούτε κάναμε κάποιο είδου επαφή και ανακοίνωση. Τα λαμβάνουμε υπόψη, με προσοχή ακούσαμε τους αναφέροντες και την διοίκηση Οπότε πρόκειται να επικοινωνήσουμε εγγράφος μαζί τους όσον αφορά τους ισχυρισμούς της αναφοράς. Thank you very much. And... Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω να πω ότι έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορέσετε να καταρτήσετε κάποιο έργο που να τα καλύπτει όλα αυτά. Πρόκειται για απόφαση των συντονιστών, που στην ημερησία διάταξη. Ε, τέλος πάντων. Για να πάμε τώρα να δούμε τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Πρώτος ο κύριος Μάτο και κατόπιν ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ που πιέζεται πάρα πολύ από το χρόνο καμιά φορά. Ακόμα και αν είναι αναπληρωτής πρώτα ο κύριος Μάτο. Δεν ξέρω, ε, αν ο κύριο ότι αλλά παίρνω εγώ το λόγο πρώτο γιατί θα, θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ του αναφέροντε. συμφωνω με, αλλά θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι όντως δεν πρόλαβε η Επιτροπή. Το είπαμε τον Ιούλιο, το ενέκρινε οι, οι συντονιστές βάλαν την προπόθεση που δεν τηρήθηκε και να, να τα τώρα. Είναι πέρα από τα νησιά όπως είπαν όλοι. Θα πρέπει να σώσουμε αυτά τα νησιά. Όλα. το είμαι από τη Λαπάλμα. Εκεί είναι τα παιδιά μου. Εκεί ζω. Φυσικά και θέλω να σωθεί το νησί. Για τι πράγμα μιλάμε. Συμφωνώ για το πώς υπάρχουν τα νησιά, αλλά δεν συμφωνώ για όλα τα υπόλοιπα. Τι όραμα έχει η Επιτροπή, τι θέλουν αυτές οι αναφορές. Θέλουν να μην παρέμβει στο κινητικό δίκαιο και θέλουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ούτε ένα επιχείρημα δεν ακούσαμε το οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχει παραβίαση ε, του κοινωτικού δικαίου μεταξύ άλλων διότι το μόνο το οποίο λέει αυτή η νομοθεσία είναι προβλέπει κάποια μέτρα, τίποτα άλλο. Είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας. Ό,τι μέτρο το οποίο εκτελείται δυνάμει κάποιου νομοθετήματος θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Έτσι κρίνεται, αν έχουμε αντίθεση προς το κοινωτικό δίκαιο. Το μόνο όμως που λέει αυτή, αυτός ο νόμος βάζει κάποιες ε, βάσεις, γενικές αρχές, και ε, δεν είναι δυνατόν να αντιβαίνουν αυτά τα γενικά πράγματα με το κινητικό δίκαιο είναι σαν λέμε ότι επειδή κάπου κάποιο αυτοκίνητο χτύπησε κάποιον απαγορεύουμε όλα τα αυτοκίνητα άρα τίποτα δεν παραβιάζει αυτό το νομοθέτημα έχουμε κάποια σχέδια που παρέχουν εγγυήσεις και βέβαια είμαι σίγουρος ότι λόγω της βιασύνη υπάρχει κάποιο λάθος κάνουμε αναφέροντας αναφορές τους πριν υπάρξει η έγκριση του νόμου για τη γη. Μα αυτός ο νόμος βοηθάει στη διαπίστωση ότι έχουμε σύνομα μέτρα και επίσης τροποποιεί την παράγραφο 8 του, της νομοθεσίας το περιβάλλον. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει μελέτη επιπτώσεων. Βεβαίω και θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον κόσμο. Βεβαίω και θα πρέπει να είναι σύνομα όλα τα μέτρα. Και όταν κάτι δεν ε, είναι συμβατό με το κοινωνικό δίκαιο, τότε είναι παράνομο. Αλλά όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Τώρα υπάρχει μόνο αυτό το νομοθέτημα, το οποίο δεν έχετε σε αντίθεση με τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συγκρούεται με την κοινωνική νομοθεσία αυτός ο νόμος για τα πράσινα νησιά ούτε και υπάρχει κάτι για το οποίο ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Να κλείσει ένα αναφορά. Μα τι λέγανε για τις καθαρίστριες. Είναι το μόνο το συγκεκριμένο που ακούσαμε. Βεβαίω πρέπει να προστατεύσουν όλα αυτά τα υπέροχα νησιά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να προκαταλαμβάνουμε έναν νόμο που πέρασε με τόσο ευρία πλειοψηφία στο κοινοβουλίο μας. Δεν περιέχει ούτε μία διάταξη που αντιβαίνει στα της Ευρώπης. Να κλείσει αναφορά, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. Φερνάντο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη γενοδορία σας που μου δώσετε το λόγο και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί πράγματι θα πρέπει να φύγω από την Επιτροπή σας πριν ολοκληρώσω τις εργασίες σας. Όπως γνωρίζετε δεν είμαι τακτικό μέλος Επιτροπής Αναφορών αλλά είμαι μέλος της ΛΥΜΠΕ και έρχομαι που και που όπως είπε και η Πρόεδρος εδώ και με μεγάλη χαρά μάλιστα γιατί ε, το κάνω και από ε, χρέος, αίσθηση χρέος απέναντι στη ε, πατρίδα μου, τα Κανάρια. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ε, συμπατριώτες μου και άκουσα πολύ προσεκτικά τη μαρτυρία τους ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα, το τοπίο, ό,τι είπατε για την γη των Καναρίων, όπου και κατοικώ και εγώ. Θα ήθελα να στηρίξω ε, και προσωπικά και να πω ότι και οι υπόλοιποι σοσιαλιστές συνάδελφοί μου στηρίζουν την αναφορά που αφορά το νόμο για το έδαφος. Ε, γιατί, και το λέω πολύ ξεκάθαρα το 4 του 2007, διότι είναι ένας νόμος που όχι μόνο αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία στο σύνολό της από το 1999 μέχρι το 2013, αλλά ε, περιλαμβάνει και έναν γενικότερο σχεδιασμό αυτός είναι ο στόχος. Μια γενική χωρο, ένας γενικός χωροταξικός σχεδιασμός που δεν περιορίζεται στο τουριστικό σχεδιασμό και αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με τον νόμο ε, που ισχύει από το 2016, ένα χρόνο. Και δεν έχουν εφαρμοστεί βέβαια οι προβλέψεις, τα προγνωστικά ότι θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις από την άρξη ισχύει αυτού του νόμου. Γιατί ένας νόμος που όχι μόνο έχει έναν ορισμένο ε, ορισμένο πεδίο εφαρμογή, αλλά και φυσικά είναι περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή. Ε, τα τρία νησιά που έχουμε προαναφέρει και στόχος είναι να αποτραπεί η κοινωνικονομική στέρηση επειδή έχει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στον τουρισμό που γνωρίζουμε όλοι πόσο ε, έχει αποτελέσει μοχλό για την εξέλιξη της οικονομίας, για την ανάπτυξη στα Κανάρια νησιά εδώ και καιρό. Υπήρξε πράγματι ευρύτατη συνένεση κοινοβουλευτική. Οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις, ε, τα τρία, οι ε, τα τρία τοπικά, τροπικές αρχές και όλες οι αρχές των ε, τριών νησιών. Ο νόμος για το έδαφος έχει εγκριθεί από τεράστια πλειοψηφία. Η νόμοι που αντικαθιστά ήταν επίσης νόμοι που είχαν εγκριθεί σχεδόν με συνένεση, με ομοφωνία πριν από 20 χρόνια. Άρα πολλαπλασιάζει αυτός ο νόμος ε, ουσιαστικά ε, τα παραθυράκια που θα δώσουν δυνατότητες παραβίασης. de sus planeamientos urbanísticos. Esto και αυτό σίγουρα επηρεάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Και πρέπει να γίνει στρατηγική περιβαλλοντική ανάλυση, να γίνει περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Γιατί υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα που αφορά τις, ε, τα παραθυράκια που αφήνει ο νόμος 4 κάθετος 2017. Πέρα θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσετε για να προλάβετε το αεροπλάνο σας. Ε, Πέμπτη είναι σήμερα, πολλοί ταξιδεύουν. Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Μην βιαστείτε υπερβολικά. Θα συνεχίσουμε τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αρχίσουμε από το τέλος. Ε, βέβαια πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Γιατί υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός ε, με τη σχετική νομοθεσία που είναι πάρα πολύ αμφίβολη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, άρα ας μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και όσον αφορά την Επιτροπή, διαπιστώνω ότι όντως έχει πάρα πολύ δουλειά, αλλά το θέμα είναι Πόσες και ε, καταγγελίες έχουν υπάρξει. Άρα θα πρέπει να έχει προτεραιότητα όλη αυτή η υπόθεση και αυτό το τόσο σοβαρό νομοθέτημα. Και ρωτώ, η Ευρώπη κάτι προστατεύει και μια περιφερειακή διοίκηση το ακυρώνει. Μα δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αν μιλάμε για προστατευόμενο περιβάλλον του βιοσφαίρας, τι θα γίνει κάνουμε μια κερκόπορτα σε αυτή την προστασία και αρχίζουμε να χτίζουμε τι θα γίνει με τις ζώνες του Νατούρα Τόσο πλούσιο το περιβάλλον και η βιοπικιλία σε αυτά τα νησιά. Υπάρχει κάποιος λόγος αντικειμονικός που να μας οδηγήσει στο συμπεράσμα ότι πρέπει να αρχίζουμε να χτίζουμε στην Ήπεθρο. Σοκάρουν αυτές οι διαπιστώσεις. Άκουσε τι είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Βεβαίω και προστατεύονται τα νησιά. Αλλά πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Ένα και πρέπει να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ουτροπία, αρχίσει μια διαδικασία παραβίαση, παραβάση τέλο πάντων. Θα πρέπει βέβαια να γίνει μελέτη επιπτώσεων. Από ό,τι μου λένε η αρμοδιότητα για τη μελή των επιπτώσεων ανατίθεται στις τοπικές αρχές. Μα είναι δυνατόν επιτροπές της γειτονιάς να αναλαμβάνουν τέτοια πράγματα. Μα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το εργαλείο και για μας και για την Κομισιόν. Και άρα θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα πολύ αυστηρά. Δεν μπορεί να, με, να μεταβιβάζεται αυτή η αρμοδιότητα. Έχω επομένω πάρα πολλέ εμβολίε. και νομίζω ότι για όλους μας προτεραιότητα είναι η προτεραιότητα του κοινωτικού δικαίου. Άρα να μείνει ανοιχτή η αναφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει τη γνωμοδότησή της. Και όταν μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει επί των συμπερασμάτων η διοίκηση. Ευχαριστώ, Πεατρίς. Η Άντζελα. Gracias, Presidenta. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και ιδίω του συντονιστέ για την απόφαση που έλαβαν για την συμπερίληψη κατεπηγόντω αυτών των αναφορών εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ αυτό ο νόμο. Αρχικά, ε, πρέπει να πω ότι μου έκανε εντύπωση η παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη μου ερώτηση είναι πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο 16 Μαρτίου του 2016 ο Επίτροπος σε άλλη ερώτηση μου απαντάει ότι η Κομισιόν πρόσφατα έλαβε από τις Ισπανικές Αρχές το πλαίσιο της εν λόγω έρευνας. Έρευνα που μου είχατε επιβεβαιώσει ότι γίνεται μήνες πριν. Από το Μάρτιο, μάλλον όχι από πότε, από τις 16 ναι, Μαρτίου που με επιβεβαιώνετε εσείς ότι έχετε τα έγγραφα που είχατε στήσει από την κυβέρνηση των Καναρίων και την ανοιχτή έρευνα, δύσκολα μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχετε ακόμη έκθεση και δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι απάτσα μας δώσετε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Και όχι, δεν το δέχομαι. Αλλού αυτά. Το ίδιο θέλω να πω στην απάντηση της Δευτέρας Φεβρουαρίου, γιατί έχω μία μακρά σειρά ερώτα-απαντήσεων από το 16 και μετά, να γνωρίζετε ότι το ότι αν ε, κηρυχθεί ένα έργο ειδικού χαρακτήρα ή ε, πολιτισμική κληρονομιά επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές ε, οδηγίες, σχετική νόμοι της ε, Ένωσης. Πληροφορίες έχετε στη διάθεσή σας. Άρα γιατί δεν έχετε έρθει με μια απάντηση για αυτή την αναφορά. Εγώ θα ξαναγράψω στον Επίτροπο για να δω τι γίνεται τέλο πάντων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες, τους άλλους παρισταμένους και την πλατφόρμα που εκπροσωπούν. Και δυστυχώς πρέπει να πω, Δυστυχώ, γιατί δεν με ευχαριστεί καθόλου, να βλέπω για μια ακόμη φορά πόσο λίγο σεβασμό υπάρχει. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για την οικολογία κτλ. και για μέτρα για την καταπολέμηση. Και άλλο ένα δείγμα σήμερα λάβαμε για το πόσο λίγο σεβασμός δίνεται στο περιβάλλον. Βλέπουμε άλλες ωρέξεις. Ε, ε, σε ό,τι αφορά την οικοδομική ανάπτυξη. Δεν ανήκουν στη σημερινή εποχή. Πουέρτο για είδη, πετρολαϊκές επιχείρησεις κτλ. Η οδηγία για τα ύδατα παραβιάζεται. Εδώ και δεκαετίες δεν καθαρίζονται τα νερά και πέφτουν στη θάλασσα. Πάνε τα μικροάλγη και λέτε να μην τα τρώμε τα φύκια αυτά, το πρόβλημα είναι ο τουρισμός να μην πηγεί. Μα δεν είναι αυτή η λύση. Συμφωνούμε όλοι νομίζω από αυτού. και επιλέγουμε κατά το δοκούν και αλακάρτα την ομοθεσία όταν μας συμφέρει. Όχι όμω παραλυτικέ οδηγίε. Κύριε Μάτο, η αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, RED Natura, ε, αντίκτυπο Natura 2000, η πρόσβαση στην ενημέρωση προφόρηση για τα περιβαλλοντικά. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά, τα, ε, πολύ διαφορετικές οι προθεσμίες γιατί ουσιαστικά με τον νόμο αυτό έχουμε ε, φτιάξει και μία παγίδα. Να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραμείνουν αυτά όταν έχουμε να κάνουμε το περιβάλλον ε, και την τουριστική ανάπτυξη. Είναι σαν να θέλουμε τελικά να σκοτώσουμε τη Χίνα με τα χρυσά αυγά. Ο στόχο και με αυτά με την προηγούμενη εβδομάδα είναι να μην υπάρχει αυτό το προστατευτικό πλαίσιο και να μπορεί να πραγματοποιείται πολεοδομική δραστηριότητα. Αλλά να μην πω και τίποτα χειρότερο, βλάπτουμε ακόμη περισσότερο το περιβάλλον με όλα αυτά. Αυτό που ζητώ εγώ είναι να εφαρμοστεί και στρέφω στην Κομισιόν τώρα. να εφαρμοστεί αρχή της προφύλαξης, γιατί ο νόμος έχει τεθεί σε ισχύ. Τι τον κάνουμε τώρα, τον νόμο τον έχουμε και η αρχή της προφύλαξης πώς θα εφαρμοστεί εδώ, αφού πλέον έχει εφαρμοστεί, δεν υπάρχει επανόρθωση. Εγώ ελπίζω ε, να εφαρμοστεί παρόλα αυτά η αρχή της προφύλαξης και για τις ε, αναφορές ζητώ να παραμείνουν ανοιχτές και για τις δύο περιπτώσεις. Ε, ουσιαστικά τις αντιμετωπίζουμε από κοινού αυτές τις αναφορές, δηλαδή όχι να κλείσουμε π.χ. αυτή για τα πράσινα και να αφήσουμε ανοιχτή αυτή για το νόμο για το έδαφος. Και οι δύο πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και θα πρέπει ε, να διαβαστούν στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, να τι μελετήσουν και εκεί, ιδίω ό,τι αφορά τι ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και περιμένω, περιμένω την απάντηση τη Επιτροπή για να τα επανεξετάσουμε τα θέματα, να μα δώσει επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Αναφορών αλλά και στου καταγγέλλοντε επιτέλου πια μια έγγραφη απάντηση, αναλυτική, διεξοδική για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. 500 έχουμε καταγγελίες και άλλες 500, το λέω ε, και το λέει και η Επίτροπος. Αλλά οι καταγγέλλοντες δεν ε, παίρνουν πληροφορίες για το πώς πηγαίνει η περίπτωση υπόθεσή τους, άρα δεν κάνουμε τη δουλειά μας αναφορές που έχουμε συζητηθεί για τα Κανάρια καλό θα ήταν να ομαδοποιηθούν. Αυτές που συζητήσαμε σήμερα, για την τεχύτητα, το ξενοδοχειακό συγκρότημα, για την κρέμη ψηλιστά στη Βερτεβεντούρα, το ε, λιμάνι Γρανδία και όλα τα άλλα θέματα που αυτά τα Κανάρια. Και κάποια στιγμή να πάμε εκεί με μια αποστολή στα Κανάρια για να δούμε τι γίνεται στις ε, ζώνε αυτές που υποτίθεται ότι είναι προστατευόμενε από το δίκτυο Natura 2000 και να δούμε τα πράγματα επιτόπου και να έχουμε τι επαφέ μα. για να δούμε και που πέφτουν αυτά τα λύματα χωρίς να έχουν καθαριστεί. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Άντζελα. Η κυρία Στανόκα, Τατιάνα, παρακαλώ. Thank you. So, on behalf of Green Zephyr Group, I want... Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά του αναφέροντες για πολύ πλήρη περιγραφή του προβλήματος. Ακούγοντάς σα, Φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης του περιβαλλοντικού ευρωπαϊκού νόμου και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγηση της νέας περιφερειακής νομοθεσίας ε, για ε, το έδαφος ε, και για τα πράσινα νησιά. Τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκα δύο φορές στην Ισπανία σε διερευνητικές αποστολές. Τη μία φορά στη Γαλλικία και μία φορά στους ποταμούς Τάχο και Εύρο που είχε να κάνει με την λειψίδρια. διαπιστώσαμε ότι όλα τα προβλήματα που έθιξαν οι αναφέροντες ήταν πραγματικά προβλήματα και πολύ σοβαρά προβλήματα. Η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να αφήσει ανοιχτές αυτές τις αναφορές και να ασχοληθεί σοβαρά με αυτές, ενδεχομένως οργανώνοντας ε, περαιτέρω αποστολές. Καταρχάς όμως θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως υπόθηκε ήδη, να γίνει σωστή αξιολόγηση αυτής της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την ε, οδηγία για τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ε, την οδηγία για τα πτηνά, για τα οικοσυστήματα κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τατιάνα. Η κυρία Εύη, παρακαλώ, Ελεονάρα. Και εγώ θέλω να έρθω και να υποστήξω τους αναφέροντες. Συμφωνώ με την αναφορά τους. Ήδη συνάδελφοι τα είπαν όλα, αλλά επαναλαμβάνω. Τα βασικά. Να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ σε σχέση με αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχών. Πρόκειται για σοβαρή απειλή για αυτό το υπέροχο περιβάλλον το οποίο πρέπει να προστατευτεί. Θα πρέπει να υπάρξει προστασία για πάντα. Έχουμε όλες αυτές τις εκστρατείες συλλογής υπογραφών. People for Soil και άλλες πρωτοβουλίες. Άρα, οι πολίτες θέλουν την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου και να μην υπάρχει αυτή η τσιμεντοποίηση χαλήνωτη οικοδόμηση. Θα πρέπει όλες οι αρχές σε κάθε επίπεδο να προστατεύουν το περιβάλλον. Ευρώπη, εθνικές αρχές, τοπικές, οπότε θα πρέπει να αποτρέψουμε εγκαίρως τις ε, απειλές από την κερδοσκοπία. Άρα, να μελετήσουμε εις τα πράγματα, να δούμε αν υπάρχει παραβίαση του δικαίου, όλα αυτά τα οποία ισχυρίστηκαν με πληρότητα οι αναφέροντες. Τι γίνεται με το στρατηγικά νομοθετήματα, την περιβαλλοντική νομοθεσία, όλα αυτά τα οποία δεν μπορεί να τίθενται να αμφιβόλω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ελεονόρα κύριος Μπενίτο Ζιλνάγκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ στις Βρυξέλλες. Σχετίζονται άμεσα αυτά τα δύο θέματα μεταξύ τους. Το ένα έχει να κάνει με το τουριστικό μοντέλο, απέναντι σε ένα πιο βιώσιμο και εφόρο τουρισμό, πιο φυσικό, σε σχέση με το τοπικό έδαφος που θα είναι ο βέλτιστος και ο πλέον αποφελής για τις τοπικές οικονομίες κάτι το οποίο προσπαθούν να εφαρμόσουν πολλές περιοχές απέναντι σε ένα μοντέλο μαζικού τουρισμού που δεν έχει σχέση με την πρόσπιση του οικοσυστήματος και την ε, τοπική οικονομία. Αυτός ο τουρισμός επίσης έχει και ένα άλλο πρόβλημα, ακόμη μεγαλύτερο, που είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να πω, είναι ότι αντιβαίνει και στην νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για μια ακόμη φορά λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια απόπειρα στην προκειμένη περίπτωση από την Ισπανική κυβέρνηση, μάλλον την κυβέρνηση των Καναρίων, να, να ε, κάνει πιο λιγότερο δεσμευτική την νομοθεσία για τα κερδοσκοπικά συμφέροντα κάποιων που θέλουν να παίξουν με το έδαφος, ε, με το περιβάλλον παραβιάζοντας ε, τους ισπανικούς ε, και ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ. Και ουσιαστικά στόχος είναι να ανοίξει πόρτα σε αυτές τις κατεπίρουσες διαδικασίες όπως υπόθηκε απορρίθμιση δηλαδή και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ε, τοπικός, ε, περιφερειακός. Και απ' την άλλη επιβάλλονται και πολύ πιο σύντομες προθεσμίες εκτέλεσης για να μην μπορεί να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Και υπάρχουν και απλουστευμένα συστήματα εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου που αντιβαίνει στην αρχή της προφύλαξης όπως είπαμε και πάνε και προλαλήσαντες. Ο κίνδυνο με όλα αυτά ποιο είναι. Να φτάσουμε, ελπίζουμε όχι βέβαια, αλλά για μια ακόμη φορά στο να φτάσουμε σε μια πολιτική τετελεσμένων γεγονότων. Και έτσι να θέσουμε σε κίνδυνο προστατευμένε περιοχές με αυτά τα νομικά τεχνάσματα, τα κολλήματα και τελικά τι θα γίνει. Η ζημιά να έχει γίνει και να είναι πολύ δύσκολο να αναστραφεί γιατί τα σχέδια προχωρούν σιγά σιγά. Δεν μπορεί να βρεθεί κανένα επιχείρημα υπέρ του κλεισίματος των αναφόρων, ιδίως από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much. now I have only one more speaker. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μόνο η κυρία Μπιλπάου απομένει στο κατάλογο των ομιλητών. Yo intervengo δεν είμαι τακτικό μέλο. αλλά που και που έρχομαι όταν υπάρχουν θέματα που με καίνε. Που με καίνε και συναισθηματικά, αλλά και πολιτικά, γιατί ξέρετε, ε, έχω στρατευθεί με τον συνασπισμό Ευρώπη του, των Καναρίων. Με αυτή την παράταξη εξελέγει. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσω τους ε, αναφέροντες πρώτα-πρώτα. Εμπιστεύομαι 100% τις περιφερειακές αρχές των Καναρίων και τα κόμματα των ε, Καναρίων. Ήμουνα στις ζητήσεις αυτές και έτσι έγινε. Τα ψήφισαν όλα αυτά. Και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι πρώτα-πρώτα υπάρχει προβληματισμό, υπάρχει μέρημνα για την προστασία του περιβάλλοντος των νήσων και άλλη μέρημνα που έχουν είναι όπως ε, είπε η Αντιπρόεδρος να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργούν θέσεις εργασίας νέες. Γιατί κάποιος από τους αναφερόντες είπε ότι σε κάποιο νησί έχουμε 25% ανεργία προστασία από τη μια και από την άλλη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα εργαστήριο τεχνολογία στο Γέρο. Είναι υδροαιολικό. Αυτό είναι σημείο αναφορά για τα νησιά και είναι παράδειγμα προς μίμηση διεθνώς. Να, τι θέλουν να κάνουν, τι θέλουν να αναπτύξουν οι τοπικέ αρχέ. Τώρα, όσον αφορά τους νόμου πρώτα το νομοθέτημα για τα πράσινα νησιά, ε, αυτό ψηφίστηκε από 80% από όλες τις δημοτικές αρχές και από όλα τα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θεμητή αυτή η διοικητική πράξη. 80% ήταν η ψήφη που συγκέντρωσε η τέτοια απόφαση δεν επιδέχεται να λέμε βλακίες. Έχει το 100% της εμπιστοσύνη μου η δική περιφερειακή αρχή. Είπαμε μέρη να είναι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά για τον νόμο που το 80% από τα κόμματα και από τις δημοτικές αρχές. Επομένως, σέβομαι τον νόμο και στρίζω τις αρχές. Δεύτερον, νομίζω ότι εδώ όπως και παντού υπάρχουν δύο πολιτικά οράματα. Αντίθετα. Όμως η πλειοψηφία πήγε προς τη μία κατεύθυνση με το 80% και τα πολιτικά κόμματα Τώρα όσον αφορά το νόμο για τη γη. Ε, και εδώ είδαμε και διαπιστώσαμε ότι είναι δέσμε μέτρων αυτή, αυτό το νομοθέτημα με το άλλο. Όταν επομένως υπευλήθη αυτή η αναφορά, η, αυτός ο νόμος ήταν νομοσχέδιο. Ε, γι' αυτό θα ήταν σωστό να δούμε τι μορφή πήρε ο νόμος. Και ακούσαμε τις εξηγήσεις της Αντιπροέδρου. Διάβασα τα σχετικά έγγραφα και άκουσα τι ελέγχθη για τα, το περιβάλλοντος, για τη συμμετοχή. Μα υπάρχουν εγγύσει προς τα επιθυμητά. Κανείς άλλος δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για την προστασία των νήσων από τις ε, περιφερειακές αρχές των Καναρίων. Ε, γι' αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να ακούγαμε την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα το μάθουμε κάποια στιγμή ποια είναι. Άρα συμφωνώ με τις περιφερειακές αρχές και θεωρώ ότι πρέπει οι αναφορές να τεθούν στο αρχείο. Ευχαριστώ πολύ. Εφόσον ήδη μακρηγόρησαν, θα έλεγα κιόλα, ε, όχι μόνο μίλησαν οι, αναφέροντες, ε, οι αναφέροντες, καλό θα ήταν να πάρουν το λόγο ένας ή δύο από εσά, όχι όλοι σας, ένας ίσως, και να είσαστε πολύ σύντομοι. Μπορώ να σας εμπιστευτώ. Ποιος θα πάρει το λόγο. Ωραία, παρακαλώ. Θυμηθείτε μόνο τι είπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με κάθε συμφωνώ στα πολιτικά κόμματα θέλω να πω ότι σέβομαι περισσότερο από τα κόμματα το κράτος δικαίου. Πρόκειται εδώ για ενιαία δέσμη μέτρων. Και θα πρέπει να δούμε ότι τώρα γίνεται μια επανάσταση στην νομοθεσία και σας παραπέμπω στα όσα είπαμε και σας ερωτώ εάν έχουμε μια τέτοια ευρεία πλειοψηφία που ενέκρινε αυτό το νόμο και στο αρχιπέλαγος είναι όλα προστατευμένα. Γιατί να γίνει αυτός ο, αυτό το αυτή δέσμη μέτρων που τα αλλάζει όλα. Και από την άλλη μεριά ξέρετε ότι είχαμε νόμους που μοιάζουν με τον νόμο για το έδαφος, για, το, για τη γη, παρόμοιες που ακυρώθηκαν από το νοτοδικαστήριο να σας δώσουμε μια έκθεση που έχουμε και που επίσης εκεί φύγονται τα θέματα νομιμότητας και αντισυνταγματικότητας. Και αυτό προέρχεται από επίσημο όργανο των περιφερειακών έργων που εξετάζει αυτά τα κριτήρια. Δεν υπάρχει εκεί αποκλειστική αρμοδιότητα. Κυριαρχεί το κοινοτικό δίκαιο. Οπότε σέβομαι τις αρχές αλλά κυρίως το κράτος δικαίου και τώρα θα τεθεί σε ισχύ αυτός ο νέος κώδικας. Παρακαλώ να την κρατήσετε ανοιχτή την αναφορά. Θα πρέπει ε, όπως επιτάσσει η δημοκρατία να γίνει σεβαστή γνώμη και της μειοψηφίας. Υπάρχει χρόνος με νυφαλιότητα εις βάθος να δούμε γιατί γίνεται όλη αυτή η απορρίθμιση του νόμου για τη γη που καταφέρεται κατά της νομοθεσίας που ισχύει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ο λεγόμενος τουριστικός νόμος για τα πράσινα νησιά που δεν είναι παρά ένας νόμος για τα γκρίζα νησιά ουσιαστικά 2 του 2016 που εγκρίθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο από το Κοινοβούλιο των Καναρίων εγκρίθηκε χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών ε, της κοινή γνώμης για τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον όπως λέει η Οδηγία 2003 κάθετος 35. Έλεγε ο Γαμπριέλ Μάτο επίσης ότι κάθε project ε, θα εκτιμηθεί με περιβαλλοντική μελέτη στρατηγικού χαρακτήρα. Δεν ε, θα γίνουν με αυστήρες προδιαγραφές αυτά τα σχέδια. Δηλαδή θα είναι και ε, ο κριτής αλλά και ο κύριος του έργου ουσιαστικά οι αρχές εκεί. Όπως έλεγε ο σύντροφος, ε, λέτε ότι στηρίχτηκε από το 80% μένα των πολιτικών κομμάτων. Αλλά δεν μπορεί αυτό να δώσει τιμοποίηση σε αυτόν τον νόμο. Εμεί ζητούμε να παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορές, γιατί θα δημιουργήσουν αυτά τα έργα επανόρθωτη ζημιά. Θα τα καταγγείλουμε και στη συνέχεια, γιατί παραβιάζουν πολλές οδηγίες ευρωπαϊκές. Ανεπανόρθωτε αν οι ζημιέ όμω. Και θα υπονομεύσουν το μέλλον των επόμενων γενιών που πρέπει να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα σαφείς. Είναι σαφές το μήνυμά σας. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Είμαι έτοιμη να κλείσουμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτές όλες τις αναφορές και λυπάμαι λίγο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να δώσει πιο πλήρη απάντηση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό γίνεται λόγω έλλειψης χρόνου. Ε, θα απευθυνθώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ε, ζητώ να επανέλθετε με περαιτέρω πληροφορίες αφού κάνετε τη σχετική έρευνα. Μπορείτε να μας δώσετε και σε τις πληροφορίες αυτές, δεν θα χρειαστεί ε, νέα συνεδρίαση για κάτι τέτοιο. Αφήνουμε όμως ανοιχτή την ε, αναφορά και θα αναλύσουμε τις απαντήσεις που θα μας στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, παραπέμψουμε το θέμα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ για να τους ευαισθητοποιήσουμε και για να έχουμε και σωστή απάντηση από την ΕΝΒΗ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα συνάδελφο το λόγο. Σας, ζητώ, σας ευχαριστώ όλους σας που αφήσατε το όμορφο πράσινο νησί σας για να έρθετε εδώ στις βροχερές Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε πολύ που παραβρεθήκατε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε που μας ευαισθητοποιήσατε πάνω στο θέμα αυτό. Και εγώ Προσωπικά σκέφτομαι ποιο από αυτά τα όμορφα νησιά να επισκεφτώ την επόμενη φορά. Πάντως σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σας εύχομαι καλή επιστροφή στα όμορφα νησιά σας. Εμείς συνάδελφοι προχωράμε στην επόμενη αναφορά 623 σχετικά με την προσφυγή EU Pilot ε, σχετικά με το δέλτα του ποταμού Λόπρεκατ. Ο αναφέρον είναι εδώ και σας δίνω με τα χαρά στο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ προσωπώ το Σύνδεσμο για την ε, πρόσπιση της φυσικής κληρονομιάς. Ε, και πα... Ναι, μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, προς ε, ένδειξη βασμού στην αναφέρουσα. Εσείς που θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλή σας από την άλλη πλευρά της πόρτας. Okay, fine. Thank Ευχαριστώ όλες και όλους. Σιγά σιγά παρακαλώ και ήσυχα να εγκαταλείψετε την αίθουσα για να δώσουμε το λόγο στην αναφέρουσα. Όταν νιώθετε έτοιμοι, ξεκινήστε. Όπως έλεγα λοιπόν, εκπροσωπώ το σύνδεσμο για την πρόσφαση της φυσικής κληρονομιάς, ΔΕΠΑΝΑ, και έχουμε καταθέσει μια καταγγελία για την καταπολεμία κατά παραβίαση της για τα οικοσυστήματα Το Δέλτα του Λιομπρεγάτη είναι το μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος υδροβιότοπος ε, στην ε, ε, επαρχία της Βαρκελός, τρίτος στην Καταλωνία και μεγαλύτερος υδροβιότοπος στην Ευρωπή, από δεν περιλαμβάνεται στο Ραμσάρ παρά στο ότι τη τα κριτήρια 2, 3, 4 και 7 και είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο δελταϊκό σύστημα στην Ιβηρική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της μεταναστευτικού οδού ε, των πτηνών ε, από τη, στη μετάβασή τους από την Ευρώπη στην Αφρική και πολλές φορές είναι ένας ε, δορυφός του εύρω. Αυτή είναι η σημασία του και γι' αυτό και έχει συμπεριληφθεί ε, στις περιοχές Global Important Bird Areas. Είναι σημαντικό αυτό το μέρος, είναι όμως εκεί πάρα πολλές υποδομές ε, και πάρα πολύ πληθυσμό. Δεν υπάρχει επαρκής προστατευόμενος χώρος, δεν υπάρχει καλή διαχείριση και υπάρχουν συνεχείς αναρνητικές ενέργειες και υπάρχει μείωση των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράτημα ένα της οδηγίας ε, για τα πτηνά και για τα πουλιά που φτιάχνουν τις ε, φωλιές τους ε, εκεί. Υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο που υποτίθεται ότι θα εκπονεί το, το ειδικό σχέδιο για την προστασία των φυσικών χώρων ήταν ένα αντισταθμιστικό μέτρο για τη δημιουργία του αεροπορίου, του αεροδρομίου. Δεν έχει όμως γίνει ακόμη δημοσίευσή του. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δει διάφορες εσωτερικές εκδοχές, αλλά κανένα ε, κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η τελευταία εκδοχή δεν περιλαμβάνει καμία από τις ελληνικές περιοχές που ορίζεται από το Import Bird Area 140 που είναι σημαντικές για πολλά από τα πτηνά του παραρτήματος 1. Το ειδικό σχέδιο ουσιαστικά είναι ένα πάζελ μεταξύ προστατευόμενων πυρχών, παραδοσιακών γεωργικών πυρχών και άλλων ένταση καλλιέργεια και άλλε που μπορούν να χτιστούν. Άρα πολύ δύσκολα εφαρμοστεί το σύνολο τη νομοθεσία γιατί δεν αντιστοιχεί αυτό το σχέδιο σε κάποιο γεωγραφικό ή φυσικό χώρο συγκεκριμένο και περιλαμβάνει διάφορες διαφορετικές περιοχές διαφορετικού σκοπού. Οι Ισπανικές αρχές νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουν επιστημονική τεκμηρίωση που θα επιβεβαιώνει τις αποφάσεις που έλαβαν ορίζοντας το χώρο όπως τον όρισαν, για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα τα μέτρα του ειδικού σχεδίου και του διαχειριστικού σχεδίου, λαμβάνοντας ε, υπόψη την, το κατακαιρματισμό. Επίσης αυτό το δέλτα είναι ειδική περίπτωση. Γιατί αυτή η ΖΕΠΑ 146 <laughs> είναι κατώτερη από το ΙΜΠΑ 140 από τα 3.500 εκτάρια που με ορνηθολογικά κριτήρια πληρούν τις, τις απαιτήσει για να μπουν σε αυτή την ε, ΖΕΠΑ, αυτή την ζώνη προστασίας, το 146, καλύπτονται μόνο κατά το 30%. Του ΖΕΠΑ. Αυτή η πρόταση λοιπόν περιλαμβάνει μόνο το νέο, τη νέα κήτου του ποτάμου Λεμπρεγάτα και τις εκβολές του, άρα δεν περιορίζει παρά τα δεν ρυθμίζει παρά τα ελάχιστα. Υπήρχε αυτό το σχέδιο εκτροπής του Λιομπρεγάτα και υποτίθεται πρέπει να προστατευτούν τα, τα πτηνά. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιστημονική μελέτη, γιατί χρειάζεται να αλλάξει η χάραξη αυτή τη ζώνη για το ΔΕΛΤΑ και να λάβουν υπόψη του στη χάραξη τις μελέτες που έλεγαν ότι πρέπει να επιμηκυνθεί, να επεκταθεί. Επίσης, θα πρέπει να περιλάβει τα ειδικά μέσα για την αποκατάσταση των πληθυσμών προστατευόμενων ε, ειδών πτηνών και να μην το αφήσει για το μελλοντικό σχέδιο διαχείρισης που δεν ξέρουμε πότε θα δημοσιοποιηθεί. Τέλος, ε, ο σύνδεσμό μα θέλει να τονίσω ότι πρέπει προστευόμενε περιοχέ στο Δέλτα του να γίνουν περισσότερε και να τηρηθούν οι δεσμεύσει που έχουν λάβει οι Ισπανικέ αρχέ. Ιδίω όταν βλέπουμε κατάφορη παραβίαση διαφόρων άρθρων των δύο οδηγιών για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα. Γι' αυτό ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Thank you. Excellent. Thank you. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δάνιελ Φερνάντες Κόμες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους αναφέροντες οι οποίοι ήταν ε, πάρα πολύ ενδελεχείς στα όσα μας ε, εξέφερσαν. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας καταγγελίας που μας είχε γίνει σε σχέση με την προστασία αυτής της ζώνης ειδικής προστασίας για πτηνά στο δέλτα του Λιομπρεγάτ. Προστατεύεται από το κοινωτικό δίκαιο σε σχέση με την προστασία της φύσης. Στη συνέχεια της καταγγελίας αρχίσαμε μία έρευνα. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις και τις κινήσεις των Ισπανικών αρχών διότι υπήρξαν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν για διάφορα σχέδια και έργα όπως για το ΠΡΑΤ, το αεροδρόμιο και αυτά που μας είπε τέλο πάντων η αναφέρουσα. Ακόμη δεν έχουμε λάβει επιβεβαίωση για το κατά πόσον όσα ανισταθμιστικά μέτρα προβλεπόντουσαν αν έχουν πλήρως εφαρμοστεί. Σύντομα θα σταματήσουμε την έρευνα και θα εξασφαλίσουμε να υπάρξουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και να εφαρμοστούν από τις αρχές τα όσα επιτάσσει το κοινωτικό δίκαιο. Και ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο συναδελφοί, μόνο εγώ και ο κύριος Μαριάς μείναμε. Άρα, κύριε Μαριά, θέλετε το λόγο. Would I like to take the floor on this? I... Μήπως θέλετε. Α, επιφυλάσσομαι να μιλήσω στην επόμενη αναφορά. Yeah. Okay. Uh, we have listened to you. We have... Σας ακούσαμε, ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας δίνω πάλι το λόγο εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι στην αναφορά αυτή. Δύο λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Hola, eh, perdón. Γεια σας. Καλησπέρα. Ε, εγώ θα λάβω το λόγο για να απαντήσω, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Θέλουμε να ξεκαθαριστεί για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν προκειμένου, περιορίζεται μόνο σε αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα σε σχέση με αυτά τα έργα όπως ε, το διεύνηση τέλο πάντων του αεροδρομίου. Εμείς θεωρούμε ότι τώρα έχουμε παραβίαση περιβαλλοντικών οδηγιών. Και επίσης παραβίαση της οδηγίας Habitat Chiaves. Προς τούτο έχουμε προσαγάγει τη σχετική επιστημονική τεκμηρίωση. Στο Δέλτα του Λεμπρεγάτη είπαμε ότι οι σχετικές προστατευόμενες περιοχές δεν έχουν προστατευτεί όπως επιτάσσουν οι κοινωτικές οδηγίες. Είχαμε ε, κριτήρια που επιστατεύτηκαν που δεν είναι επιστημονικά. Τα κριτήρια είχαν να κάνουν με την οικοδόμηση. Κυριάρχησαν τα συμφέροντα. Τα ξέρετε και από άλλες αναφορές. Πολλές φορές δεν κυριαρχεί το συμφέρον προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά άλλα συμφέροντα. Ούτε η καταλλανική κυβέρνηση φύρμωση τις ε, οδηγίες όσον αφορά την περιχαράκωση των προστατευομένων περιοχών. Άρα αυτό να εξεταστεί, αν γίνανε όλα επιστημονικά ή ου. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαριά, συμφωνείτε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή μέχρι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη να έχει αξιολογήσει το σχέδιο για το ΔΕΛΤΑ αυτό από τις Ισπανικές Αρχές. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κάνουμε έτσι. Θα προχωρούμε. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, που είναι η αναφορά 1389. Σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο που εκτελείται στο ρέμα της πικροδάφνης, ρέμα μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας και τις φερόμενες ως παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω είναι εδώ συνήθω. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Γιάννη Κονινιώτη. Παρακαλώ. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord vous confirmer que suite à la dernière commission... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατόπιν τη τελευταία μα ανακοινώσεως προ την Επιτροπή σα. δεν έχουμε λάβει άλλα στοιχεία για αυτό το έργο. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσον υπάρχει εδώ πέρα παραβίαση της νομοθεσίας έχει υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Νοέμβριο θα εκδικαστεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω όπως θα ξέρετε ότι η Επιτροπή ούτως ώστε να αποδώσει δράσεις υπέρ του πολίτη, έχει δώσει προτεραιότητα σε κάποιες οριζόντιες δράσεις. Θέλουμε να υπάρχει στρατηγικός αντίκτυπος. Οπότε στην πρόσφατη Ανέγκριση Επιτροπής, τη 19 πρώτου του 2017, ε, ονομάζεται Ευρωπαϊκό Δίκαιο για περισσότερα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διεκπεριώνει κάποια φακέλους, κάποια θέματα ε, που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και έτσι συνδέονται με άλλα θέματα. Οπότε φαίνεται τώρα η πρόκληση που έχει εντοπίσει η Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων της ε, πλημμύρας. Γιατί ε, το είπε αυτό ο αναφέρον, ότι με αυτό το έργο κινδυνεύει περισσότερο τώρα η περιοχή από τις πλημμύρες Οπότε και αρχίσαμε δύο διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδος. Και έτσι θεωρούμε ότι η οδηγία 60 του 7 ε, που αφορά τις ε, πλημμύρες θα εφαρμοστεί. Έχουμε επίσης το, το, το, το φάκελο 71 που αφορά αυτές τις ζώνες που επιδέχονται κίνδυνο πλημμύρας και υπάρχει το σχετικό πλάνο, σχετικός χάρτης και η Ελλάδα πρόσφατα ε, μας έδωσε τα στοιχεία που θέλουν σχετικούς χάρτες, οπότε και εμείς ε, προχωρήσαμε στην αρχιοθέτηση της προσφυγής για παραβίαση. Τώρα, όσον αφορά την ε, δεύτερη προσφυγή, έχουμε την, την έγκριση αυτών των σχεδίων προστασίας από τη τις πλημμύρες. Εδώ πέρα έχουμε πάλι το θέμα της οδηγίας, τόσο ώστε να γίνεται σωστή αξιολόγηση αλλά και άρτια προστασία του εδάφους από την ε, πλημμύρα. Ε, εμείς στις 28 Τετάρτου του 2017 απευθύνουμε προειδοποιητική ε, επιστολή και έχουμε λάβει την απάντηση. Προσπαθούμε επομένω να βοηθήσουμε τις εθνικές, ελληνικές αρχές όχι μόνο με την διαδικασία επί δηλαδή με τον μπαστούν και με τον καρότο. Απλώ θέλουμε να κάνουμε και διμερεί επαφέ. Και σε μία συνάντηση που θα γίνει τέλειο Οκτωβρίου στην Ελλάδα θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε τα πιο σημαντικά που έχουν σχέση με αυτή την ε, παράβαση του δικαίου. Και έχουμε όλες αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν σχέση με την αναφορά. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη κάθε φορά που γίνεται αξιολόγηση αυτού του προγράμματος που θα πρέπει να εγκρίνει ε, και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή ε, η Ελλάδα για την περιοχή της Αττικής. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Ήρθε η ώρα. Η ώρα σας. I don't think so. Uh, θέλω να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα είναι μια σοβαρή καταγγελία που έχει γίνει από πλευρά των αναφερόντων. Δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σήμερα. Ε, όμως είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν στους ισχυρισμούς της ε, Κομισιόν με έγγραφο το οποίο έστειλαν και το οποίο υπάρχει μέσα στο ενημερωτικό που έχουμε ως ε, Ευρωβουλευτές. Το δεύτερο θέμα είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με το ρέμα της πικροδάφνης διότι έτσι όπως ε, έχουν ε, ρυθμιστεί τα πράγματα, στην ουσία αντί να αποτελεί ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα βοηθούσε στην ε, περίπτωση αυτή, έχει εξελιχθεί σε ένα τρομερό πρόβλημα για σημαντικές περιοχές στην Αθήνα, όπως είναι η Λιούπολη, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλυμος και το Παλαιό Φάλιρο. Επομένως το βασικό που αναφέρουν οι καταγγέλλοντες ε, και που επιμένουν είναι ότι αντί να έχουμε μία ρύθμιση αντιπλημμυρική, επί του πρακτέου έχουμε μία παραβίαση ουσιαστικά της ίδιας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και αντίθετα αποτελέσματα. Επομένως η Κομισιόν θεωρούμε ότι έχει αρμοδιότητα διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι ένα έργο σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει όλες οι πλευρές ενός έργου να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για να βλέπουμε αν υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Νομίζω ότι η αναφορά είναι πλήρης ως προς τα επιχειρήματά της και ε, οπωσδήποτε δίνει την ευκαιρία στην Κομισιόν αν θέλει να παρέμβει, να παρέμβει. Ουσιαστικά το είπε λίγος πολύ η Κομισιόν. Τι είπε ότι το γενικό πλαίσιο και η εφαρμογή της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ελλάδα πάσχει. Επί της ουσίας έχει πάρει μέτρα και μάλλον θα οδηγηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Επομένως θα έλεγα ότι έμεσα αναγνωρίζει ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία είναι, η αναφορά είναι πραγματική, έχει βάση και θα πρέπει να ασκηθεί πίεση ώστε να ρυθμιστούν ε, τα θέματα αυτά. Το ότι η υπόθεση έχει πάει στο Συμβούλιο Επικρατεία θα έλεγα ότι έχει και επιβοηθητικά στοιχεία. Δηλαδή ούτω ή άλλω θα βγει μια απόφαση από το ελληνικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν αποτρέπει εμά εδώ ω Επιτροπή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, να δώσουμε απαντήσει στου αναφέροντες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η αναφορά οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Θα πρέπει η Κομισιόν να λάβει υπόψη τα επιχειρήματα που απέστειλαν ε, το τελευταίο διάστημα οι ίδιοι οι αναφέροντες και να δει ξανά όλα τα επιχειρήματά τους, γιατί είναι αρκετά τα επιχειρήματα που στηρίζουν την ε, αναφορά. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια επιστολή στην περιφέρεια Αττικής για το θέμα αυτό, στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ε, Δημοσίων Έργων, ας το πούμε, ε, που είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Τέλος, το σοβαρό ζήτημα του πώς αντιμετωπίζονται οι πλημμύρες νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Πρέπει να είναι με τρόπο που εφαρμόζεται η ίδια η νομοθεσία. Ε, αυτά κυρία Πρόεδρε. Φαντάζομαι τώρα βλέπω και οι συνάδελφοι οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν έρθει. Θα ακούσουμε και τις απόψεις των συναδέλφων και επιφυλάσσουμε αφού ακούσουμε την απάντηση της Κομισιόν να προσθέσω αν χρειαστεί κάτι στη συζήτησή μας και φυσικά να ακούσουμε την πρότασή σας για το πώς θα χειριστούμε την υπόθεση. Ευχαριστώ. Mrs. Κυρία Σακοράφα. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα ε, το αργά το απόγευμα, αλλά παρόλα αυτά καλώ ήρθατε. Ε, οι αναφέροντες στη συγκεκριμένη αναφορά μας καταγγέλνουν ότι στο συγχρηματοδοτούμενο έργο, κυρία Πρόεδρε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εκτελείται σε ρέμα της Αττικής, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πικροδάφνης και περιλαμβάνει αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις μετά τις πυρκαγιές του 1998, υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ενωσιακής νομοθεσίας λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ασυμβατότητες με τους κανόνες χρηματοδότηση από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και απουσίας διαβούλευση Κυρίω κυρίως αυτό από τους πολίτες. Θεωρώ ότι τις καταγγελίε τους αυτές τι έχουν τεκμηριώσει συγκεκριμένοι πολίτες πλήρω και με την αφορά και τα συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία έχουν προσκομίσει. Ε, σύμφωνα όμω με τα συνημμένα έγγραφα της Επιτροπής, η οποία μας απαντά ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν παράβαση των αφαιρεμένων οδηγιών, ε, μας ενημερώνει η Επιτροπή ότι βάσει τη οδηγία 2007 κάθετο 60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρα, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταρτήσουν χάρτες επικίνδυνότητα πλημμύρα και χάρτες κινδύνων πλημμύρα, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα σε επίπεδο περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή μονάδας διαχείριση, όπω αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφο 2 συνημένο β καθώ και να καταρτήσουν σχέδια διαχείριση κινδύνων πλημμύρα που συντονίζονται στο επίπεδο τη περιοχή Λεκάνη, απορροή ποταμού ή τη μονάδα διαχείριση, όπω αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφο 2, στοιχείο Β. Οι υποχρεώσει αυτέ θεσπίζονται αντιστοίχω στα άρθρα 6 και 7 τη οδηγία με στόχο την κατάρτιση, όπω απαιτείται από το άρθρο 1 πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρα, με στόχο την μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τι πλημμύρε στην Ένωση. Δεδομένου λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν έχει εκπονήσει του χάρτε και τα σχέδια που απαιτούνται, η Επιτροπή αποφάσισε να ανοίξει έναν φάκελο επί παραβάση για κάθε ένα από αυτά τα θέματα, έναν το 2015 για την έλλειψη των χαρτών και έναν φέτο για την έλλειψη των σχεδίων. Εφόσον λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν έχουν καταρτιστεί οι χάρτε επικινδυνότητα πλημμύρα, θα ήθελα να επισημάνω στην Επιτροπή ότι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη στην αναφορά στον κίνδυνο πλημμύρα που έχουν καταθέσει με την επιστημονική του ιδιότητα μία χημικό περιβαλλοντολόγο, επιθεωρήτρια περιβάλλοντο και μία πολιτικό-Μηχανικό και γεωλόγος και μία περιβαλλοντολόγο. Συγκεκριμένα λοιπόν οι κυρίε αυτέ αναφέρουν ότι οι ποσότητε του νερού που θα εισρεύσουν στην πικροδάφνη εάν οι εργασίε αποπερατωθούν υπερβαίνουν αυτέ που το ίδιο το ρεύμα έχει δυνατότητα να αντέξει ω ε, φυσικό ρεύμα. Περισσότερα αυτά νερά θα διαβρώσουν τα, τα τη στη λοφόρη τη Βουλιαγμένη έως την εγκολή και θα διαταράξουν το φυσικό ανάγλυφο του οικοσυστήματος μαζί με την κάθε μορφή σχλωρίδα και πανίδα με αποτέλεσμα να προκληθεί ανατροπή τη ισορροπία του τοπίου. Και βεβαίω αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιώδη υποβάθμιση του υδατορέμματο και κυρίω πλημμυρικά φαινόμενα στι παραρεμάτιες περιοχέ, οι οποίε και λόγω τη θέση του έχουν ήδη χαρακτηριστεί από το ΠΚΑ, από τη Γενική Γραμματεία δηλαδή των Ιδάτων, αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου. Όλα αυτά, και αυτό πρέπει να προσέξουμε κυρία Πρόεδρε, έχουν σαν συνέπεια να ταθεί σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας των πολιτών. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να κρατηθεί ανοιχτή η, η αναφορά ε, και, να, να ε, και να, έχει ενημέρωση από τις αρμόδιες ε, εθνικές αρχές πάνω στο θέμα. Αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαι βέβαια μέλος της Επιτροπής Αναφορών. Έχω μια προηγούμενη θητεία και ισχυρίζομαι και μια τριβή με τα θέματα αυτά και επομένως την επιχειρηματολογία μου όπου αναφέρομαι σε οδηγίες δεν θα κάνω εκτεταμένη παρουσίαση, θα τις επικαλεστώ αθρηστικά προκειμένου να υποστηρίξω την αναφορά. Υποστηρίζω λοιπόν την αναφορά των κατοίκων που συζητάτε εδώ διότι πρόκειται πραγματικά για ένα έργο που έχει άμεσο και μεγάλο κίνδυνο προς το περιβάλλον και γιατί έχουμε κατασπατάληση και οικονομικών και φυσικών πόρων. Επομένως, η Επιτροπή μας μπορεί να το συζητήσει βεβαίως, έχοντας εμπιστοσύνη και στην ευαισθησία μας και στην ευαισθησία αυτής της Επιτροπής για τέτοια θέματα. Ε, το έχετε δει, την έχετε δει την αναφορά αναλυτικά, έχει κατατεθεί από το 2015. Έχετε και τα πρόσθετα στοιχεία, δεν θα τα επικαλεστώ, ξαναλέω αναλυτικά, ε, αν χρειαστεί στη συνέχεια της συζήτησης. Έχετε ακούσει τους ισχυρισμούς της Κομισιόν. Δυστυχώς δεν άκουσα τη σημερινή τοποθέτηση των κυρίων, ε, του, του κυρίου, του προσώπου της Κομισιόν και επομένως αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση, αν έχουμε διαφορετική γνώμη στη συνέχεια, το λέω. Η πρώτη μου όμως παρατήρηση για τις μέχρι τώρα απαντήσεις που δίνει η Κομισιόν στις αιτιάσεις των κατοίκων σχετικά με το θέμα αυτό ε, νομίζω ε, χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, δεν είναι τεκμηριωμένες. Μάλιστα οι εξηγήσει που δίνει σε ορισμένα σημεία ουσιαστικά φάσκουν και αντισφάσκουν παράγραφο με παράγραφο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, απλώς κάνω αυτή την παρατήρηση για να πω στο τέλος το τι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Η Κομισιόν πρέπει να δίνει πιο εμπεριστατωμένες, πιο τεκμηριωμένες απαντήσεις και να ακούει πιο σοβαρά τις αιτιάσεις που αναφέρονται στην, ε, στην αναφορά και τις οποίες εντάχει επειδή ακούστηκαν και άλλες απόψεις για να μην ε, τα ίδια πράγματα θέλω να πω ότι υποστηρίζω την αναφορά και είναι δικαιολογημένο το αίτημα των κατοίκων για τους εξής λόγους. Το πρώτο ότι παρανόμως το έργο έχει απαλλαγή ότι το έργο έχει παρανόμως απαλλαγή από περιβαλλοντική, περιβαλλοντική αδειοδότηση αφού στην οδηγία 2092 του 2011 στο άρθρο 4,4 ε, παράγραφος 3 προβλέπει ρητά ότι απαιτείται σε περίπτωση υγροτόπων περίπτωση που ισχύει για το ρέμα πικροδάφνης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εδώ είναι και οι αντιφάσει τη Επιτροπή στι σχετικέ απαντήσει. Αυτή είναι η νήξη στο θέμα αυτό. Δεύτερο, το έργο δεν γνωστοποιήθηκε στο κοινό δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν μεταξύ ενός Δήμου και της Περιφέρειας παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την οδηγία την ίδια την 92 του 2011 στο παρακάτω άρθρο, στην παρακάτω παράγραφο, καθώς επίσης παραβίασε και τις συνθήκες του άρχους, η οποία είναι γνωστή στην ε, Επιτροπή μας. Δεν θα ε, ε, αναλύσω περισσότερο τι σημαίνει αυτό. Τρίτος λόγος το έργο παραβιάζει την οδηγία, του στόχου, συγγνώμη, τους στόχους των οδηγιών 60 του 2000 και 60 του 2007 αφού δεν έχει εκτιμηθεί και δεν έχει αξιολογηθεί δεόντως ο κίνδυνος πλημμύρας μέσω σχετικής μελέτης. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο, ε, διότι ε, δεν έχει εκτιμηθεί σωστά ο περιβαλλοντικός κίνδυνος και ο κίνδυνος πλημμύρας, και επομένως η αναγκαιότητα των έργων προκύπτει από αυτό, ενώ στην ουσία το έργο δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους για πλημμύρα στην υφιστάμενη απορροή των, νερών από τους δύο αγωγούς στο υφιστάμενο ε, ρέμα της πικροδάφνης. Τέταρτο, δεν αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι πλημμυρών, ίσα ίσα τριπλασιάζονται, αυτό που προσπαθώ τώρα να αναλύσω, καθώς ενσωματώνεται τα ύδατα από δύο αγωγούς που δεν ανήκουν στην ίδια λεκάνη με το υφιστάμενο ρεύμα και αυτό επιβεβαιώνεται από τρεις επιστήμονες με διαφορετικές ειδικότητες Αναφέρθηκε συνάδελφο Σακοράφα, δεν θα επεκταθώ και εγώ σε αυτό. Πέμπτο, το έργο θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση των άγριων πτηνών, παραβιάζοντας την οδηγία 147 του 2009. Έκτο, παραβιάζει την αρχή αναλογικότητα κατά την ανάλυση που έκανα πριν δεν αντιμετωπίζεται ο, κίνδυνος πλημμύρας με αυτά τα μέτρα, αντιστρόφως ε, με τα μέτρα αυτά, δηλαδή με τη ε, ε, διενέργεια του έργου, πολλαπλασιάζεται κατά την άποψή μου και κατά τον ισχυρισμό των αναφερόντων. Έβδομο και σημαντικότερο και τελευταίο, για να μην σας κουράζω όπως υποσχέθηκα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αναγνωρίσει αρχικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, αυτούς που εγείρει η ένσταση, έχει διατάξει την προσωρινή διακοπή των έργων, η απόρριψη της προσφυγής στη συνέχεια έχει γίνει λόγω εκπορθέσμου και όχι επί της ουσίας. Κατόπιν τούτου λοιπόν ε, προτείνω αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρος, η Επιτροπή πρώτον να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά, δεύτερο να ε, συστήσει την άμεση αναστολή των έργων που γίνονται, για τα άλλα έργα στη συνέχεια ήδη έχει μπει φραγμός. Έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ένα από τα προβλήματα που έχει αυτό το έργο είναι ότι ε, έχει σαλαμοποιηθεί αυτό το, το θέμα και επομένω οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την διεξαγωγή του, αυτών των έργων που συνεχίζονται ε, ε, υφίστανται και επομένω χρειάζεται άμεση αναστολή και σε κάθε περίπτωση και τελειώνω η δική μα η απόφαση θα πρέπει βεβαίω να ζητάει περισσότερε πληροφορίε και διευκρινήσει και από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντο και βεβαίω από την Κομισιόν να απαντήσει τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα στι αιτιάσει. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Okay, colleague. Συνάδελφοι, θα κάνουμε ω Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα ζητήσουμε πολύ πιο πλήρεις έρευνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στείλουμε επιστολή στην Περιφέρεια Αττικής και στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και υποδομών. Για να ρωτήσουμε πώς έχει η κατάσταση και για να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους ισχυρισμούς των αναφερόντων. Να δούμε τι έχουν να πούν και πώς μπορούν να απαντήσουν. Και τέλος, θα ζητήσουμε πλήρη επισκόπηση του έργου, διότι αυτό λείπει. Ε, διάφορα κομματάκια μαθαίνουμε. Μία τελευταία πληροφορία από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι ότι εκρεμεί η υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο και ε, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία 15 Νοεμβρίου. Ε, όταν λοιπόν έχουμε εκρεμούσα δικαστική ε, διαδικασία, περιμένουμε και παρακολουθούμε. Όταν υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε το θέμα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά βλέπω τον κύριο Μαριά να μου χαμογελάει ε, ε, πάνω σε θέμα ελληνικής αναφοράς. Ε, έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Μας αξίζει μετά από την πολλή δουλειά που κάναμε σήμερα. Θα σας ξαναδώ σύντομα. Καλό σας βράδυ.